Συνάδελφοι, ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνατε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο επαριθμών 2. Δημόσια ακρόαση με την Ντανιέλ Νουή, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να σας καλωσορίσω, κυρία Ντανιέλ Νουή, να σας συγχαρώ για την πολύ σημαντική σας εργασία σε σχέση με την συνολική αξιολόγηση και τα όσα κάνετε στο εποπτικό σκέλος των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Στην ακρόαση αυτή θα συζητήσουμε ακριβώς τα αποτελέσματα της σφαιρικής αυτής αξιολόγησης, αλλά θα μας πείτε και ποια είναι τα επόμενα βήματα, η δημιουργία του ε, ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Επίσης είχαμε την τελευταία τριμηνία έκθεση για την πρόοδο και την υλοποίηση του κανονισμού για το ενιαίο εποπτικό ε, μηχανισμό που έχει μοιραστεί στα μέλη της Επιτροπής και Τώρα τον Νοέμβριο θα αναλάβει τι πλήρε εποπτικέ τη αρμοδιότητε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ιστορική η στιγμή και για την Επιτροπή μα, διότι έχουμε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία του ε, ενίου μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν δίνοντας το λόγο στην ε, κυρία Νουή και μετά θα έχουμε με πεντάλεπτη θηρίδα την φάση των ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ. Στον κύριο Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ ενώπιον σα κυριολεκτικά. Μια μέρα πριν η Κεντρική Τράπεζα ανλάβει τα υποπτήρια καθήκοντα σε σχέση με τι αποφάσει του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου χρόνου τόσο ώστε να μπορέσουμε να ε, εντείνουμε την προετοιμασία μα όσον αφορά τον νέο μηχανισμό αποπτήρια και όλο αυτό το έργο μας πρόκειται αύριο να δείξει τους καρπούς του και γι' αυτό το πιο σωστό είναι το να σας ενημερώσω τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Λαού για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει μέχρι σήμερα. Πέρυσι ήταν ε, πιθανός ε, το έτος πιο μεγάλη πρόκληση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ένας από τους βασικούς λόγους, γιατί εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τον υποπτικό μας ρόλο, ακριβώς γιατί αυτού του είδους την ε, ολοκληρωμένη ε, εκτίμηση και αξιολόγηση την έχουμε φέρει εις πέρας. Επρόκειτο για ένα check-up έλεγχο της κατάστασης της υγείας του τραπεζικού συστήματος, ώστε μπορούμε τώρα ε, να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς όλους τους οικονομικούς συνεργατές που ασχολήθηκαν και οπότε τώρα μπορείτε με αυτόν τον μηχανισμό να έχετε ε, εντελεχή ενημέρωση, κάτι το οποίο πρόκειται να πάει μπροστά την ε, εποπτεία για το άμεσο μέλλον. παρόλα αυτά όμως ε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση για το κοινό και πρόκειται για μια διαφάνεια σημαντικό στοιχείο ούτω ώστε να αποκτήσουν οι επενδυτέ ε, ε, εμπιστοσύνη στο τραπεζικό μα σύστημα. Παράλληλα με αυτό του είδου το αξιολογικό έργο τώρα επίσης έχουμε κάνει το προσκευαστικό έργο για τον ενιαίο μηχανισμό, τον SSM και είδατε τις τρίμνες εκθέσεις τις οποίες από τον περασμένο Νοέμβριο σας έχουμε υποβάλει και η τέταρτη από αυτές εκθέσεις σήμερα δημοσιοποιήθηκε, οπότε στο σύνολό τους αυτές οι εκθέσεις δείχνουν ότι η Κεντρική Τράπεζα τώρα έχει όλες τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ε, ικανότητες και δυνατότητες για τον υποπτικό της ρόλο και γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι χαρούμενοι που σας επιβεβαιώνω ότι είμαστε έτοιμοι για να αναλάβουμε την ευθύνη μας όσον αφορά την ενιαία υποπτία ε, των ε, τραπεζών της Ευρωζώνης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και εσάς να συγχαρούμε, εσάς τους συνομοθέτες οι οποίοι παίξατε έναν ε, ρόλο κλειδί για αυτό το φιλόδοξο σύστημα που κάνει πιο ασφαλές το τραπεζικό μας σύστημα και έχουμε τώρα την Τραπεζική Ένωση που εξασφαλίζει ότι το σύστημα μπορεί και πάλι να χρηματοδοτήσει την οικονομία οπότε και πάλι να κινητοποιήσει την οικονομική ε, ανάπτυξη και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε στη συρρήκνωση την υψηλού επέδου ανεργία και τώρα για να στραφούμε σε αυτές τις, αυτά που δημοσιοποίησαμε περισμένη εβδομάδα για την αξιολόγηση και να δούμε ποια είναι τα τελευταία στοιχεία ή στην προπαρασκευαστική εργασία του ενιαίου μηχανισμού τότε που αποκαλύψαμε, ε, ε, επομένως και δημοσιοποίησαμε αυτού του είδους την αξιολόγηση της 26 Οκτωβρίου. Αυτό ήταν ένα, ένα, ένα ορόσημο όσον αφορά το καινούριο καθεστώς εποπτείας ε, ή στην Ευρωζώνη. Και τώρα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά όργανα τα οποία πρόκειται να υπαχθούν στην ε, άμεση εποπτεία της σχετικής τράπεζας και τώρα είδατε πως γίνεται αυτό με ανεξάρτητο τρόπο, γίνεται με τρόπο ενδελεχή, αυστηρό και με συνέπεια και έτσι τώρα έχουμε ε, υψηλά πρότυπα και στάνταρ εποπτείας για όλο τον ενιαίο μηχανισμό. Οπότε όλοι αυτοί η, ενέργεια, όλη αυτή, αυτό το έργο το επιτελέσαμε και έτσι τώρα έχουμε μια αξιόπιστη βάση για το μέλλον, για τη συνεργασία και αυτό είναι ένα, ένα σημείο κλειδί για την επιτυχία αυτού του ενίου μηχανισμού και τέλος μπορέσαμε να έχουμε μια εκτεταμένη συνεργασία σε όλες τις μονάδες και υπηρεσίες που έχουν λάβει την εποπτεία και υπάρχει βέβαια ε, ομαδικό πνεύμα για όλο το προσωπικό μας που έχει ασχοληθεί με αυτό το έργο και τώρα να σας πω που καταλήξαμε και είναι διτό το μήνυμα πρώτα πρώτα να δούμε εάν πετύχαμε τους στόχους και δεύτερον εάν η έλλειψη ε, κεφαλαίων θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Έχουμε 130 τράπεζες οι οποίες συμμετέσχουν και έχουμε στοιχεία ενεργητικού που ανέρχονται στα 22-3 και αυτό σημαίνει το 80% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της Ευρωζώνης και υπό την εποπτεία μας είχαμε 6.000 εμπειρογνώμονες από τις ε, ε, αντίστοιχες ε, αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και τους τρίτους εμπλεκομένους σε αυτού του είδους την εκτεταμένη εποπτεία οπότε τώρα έχουμε περισσότερη εποπτεία όσον αφορά την ποιότητα και την διαφάνεια το ενεργητικό των τραπεζών είχαμε για πάνω από 800 συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια έναν έλεγχο είχαμε 119.000 ε, ε, δανειστές και πιστωτές που ανελήθησαν ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή και επίσης θέλουμε τώρα να φτάσουμε συναρμονισμένο ορισμό όσον αφορά την, την έκθεση των τραπεζών και τώρα έχουμε αυτόν τον έλεγχο του, της ποιότητας του ενεργητικού που φτάνει στα 7,5 δις ευρώ όσον αφορά τις τράπεζες για αξιόγραφα, για αξίες μέχρι 31 μέχρι 13 και όλα αυτά ε, αφορούν κάποιους προσαρμογές σε συγκεκριμένες ε, διατάξεις όσον αφορά ε, την έκθεσή τους σε συναλλαγές ούτω ούτω υπήν, οπότε τώρα έχουμε κάποιο, αυτό το συνολικό αποτέλεσμα που φτάνει σε κάποιο είδους ε, θεωρητική απογύμνωση από το κεφάλι 263 δις για έναν ορίζοντα τριετή. Οπότε όλη αυτή, όλος αυτός ο έλεγχος είδε ότι υπάρχει μια έλλειψη 24,6 δις ευρώ για 25 τράπεζες. Παρ' όλα αυτά 12 από τις τράπεζες αυτές ήδη κάλυψαν αυτή την έλλειψη διότι έκαναν αύξηση με το κεφάλι το 2014. Οι δε που τους λείπει αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να παρουσιάσουν κάποια αντίστοιχα ε, σχέδια ε, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ε, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η έλλειψη, γιατί θα, θα, ανάλογα από το πού προέρχεται υπάρχει διαφορετική προθεσμία σε σχέση με το από πού τους λείπει επομένω το κεφάλαιο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τώρα ότι ο δικό τομέα μπορεί να καλύψει μόνο κάποιε περιπτώσει που δεν υπάρχει άλλη λύση. Οπότε τότε θα ισχύσουν οι κρατικοί κανόνες και τότε θα φέρουν το βάρος και θα το μοιραστούν οι μέτοχοι και οι ε, ελάσσονες πίστοτες Πέραν αυτού, εγώ πιστεύω ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην έλλειψη κεφαλαίου τράπεζα με κάποια εσωτερικά μέτρα και με την πρόσβαση στις χρηματαγορές, οπότε έτσι θα πρόκειται να βοηθήσουμε τον ισολογισμό τους, να ίσως και ληστεί και αυτό πρόκειται να φέρει μας περισσότερη εμπιστοσύνη. Επίσης, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και πριν ολοκληρώσουμε αυτό, αυτή την, αυτόν τον έλεγχο, οι τράπεζες προσδοκούσαν βελτίωση όσον αφορά το κεφάλαιό τους. Και το front loading που έγινε όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης του ενεργητικού από τις τράπεζες οδήγησε σε περισσότερο από 200 δις ε, από τον Ιούλιο του 2013 με αυτά τα επιπλέον μέτρα. Για να δούμε τώρα τι άλλου είδους άλλες ε, και προπαρασκευαστικές έχουμε. Εμείς επομένως έχουμε εντατική προετοιμασία για αυτό το έργο μας όσον αφορά ε, την επιχειρησιακή αλλά και νομική υποδομή του μηχανισμού. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν τώρα θεσπιστεί κάποια σημαντικά νομοθετήματα του τελευταίους μήνες και έχουμε την απόφαση όσον αφορά το διαχωρισμό μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και του υποπτικού της υποτικής λειτουργίας. Επίσης έχουμε τον ε, κανονισμό όσον αφορά τα έξοδα της εποπτείας. Επίσης αρχέ του 2015 πρόκειται να εγκριθεί ο κανονισμός όσον αφορά ε, τις εκθέσεις, τις σχετικές με την εποπτεία. Ε, έγινε σχετική διαβούλευση 20 Οκτωβρίου. Το Σεπτέμβριο είχαμε τον οδηγό όσον αφορά την εποπτεία και, και επίσης για να μπορέσουμε τώρα να μελετήσουμε από κοινού τα στοιχεία κλειδί, ε, όλα τα στοιχεία τα οποία κινητοποιούν αυτό το μοντέλο της εποπτείας. Θα πρέπει να ε, έρθουμε να, να τα κοινοποιήσουμε αυτά και στον κόσμο και σε διάφορα θεσμικά όργανα, οπότε θέλουμε να έχουμε μια αρμονισμένη προσέγγιση, οριζόντια λειτουργία, γιατί ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια προσπάθεια πολυεθνική, είναι κάτι το καινοτόμο με αυτές τις, ε, τις κοινέ ομάδες από το προσωπικό μας και από τις εθνικές αρχές. Ε, οπότε, για αυτόν τον τρόπο έχουμε κινητοποιήσει 900 υπαλλήλους και στελέχη στις γενικές μας διευθύνσεις και στις ε, άλλες υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας. και άλλοι έχουν προσληφθεί αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα, θα είναι όμως και επομένως οι αρμόδιοι με τις προσλήψεις έχουν ε, λάβει σχεδόν 21.000 αιτήσει για θέσεις εργασίας σε αυτή την εποπτική λειτουργία και 3.000 ε, βοηθητικούς. Κάποιοι από τους ε, νέους υπαλλήλους πρόκειται να λάβουν τα καθηκοντά τους αργότερα και πρόκειται για 90 πρόσωπα. Και τώρα ολοκληρώνουμε αυτές τις διαδικασίες προσλήψεων α, περί τα τέλη Νοεμβρίου. Και το 2013 τότε που προγραμματίσαμε αυτού του είδους τον, ε, την ενέργεια αξιολόγηση και αρχίσαμε τον μηχανισμό της εποπτείας, θεωρήσαμε ότι δεν είναι αυτονόητο να πετύχουμε το στόχο μας. Οπότε γι' αυτό και σας λέω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω το, το Εποπτικό Συμβούλιο, το εκατοντάδες υπαλλήλους μας, επαγγελματίες, τους μάναζερ της Κεντρικής Τράπεζας, προσώπους των Εθνικών Αργών, γιατί όλοι αυτοί ακάματα δούλεψαν για μήνους, τόσο ώστε να μπορέσουμε τον ενίο μηχανισμό να τον ξεκινήσουμε ε, όπως είχε προγραμματιστεί. Από αύριο δηλαδή οπότε και τώρα και εμείς είμαστε έτοιμοι να λάβουμε το, τα καθήκοντά μας ε, και οπότε θα είμαστε όπως είπαμε, θα είμαστε πάρα πολύ ε, αυστηροί, θα είμαστε όμως δίκαιοι θα λογοδοτούμε, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε ανεξάρτητοι. Οπότε γι' αυτό σα λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η έννοια τη αυστηρή λογοδοσίας, ακριβώ όπω προβλέπει και ο κανονισμό ε, του ενίου μηχανισμού, όπω προβλέπει η Διοργανική Συμφωνία με το, το Κοινοβούλιο, όπω βλέπει το Μνημόνιο κατανόηση με το Συμβούλιο. Και σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ό,τι πιο φιλόδοξο έχει γίνει ποτέ από μια κεντρική τράπεζα, ανεξάρτητη για το εποπτικό της έργο, πιστεύουμε ότι κινούμεθα ή στα, στο, στο, πνεύμα αυτού του πλαισίου ε, εν κατακλείδη θα πρέπει να σας επαναλάβω τα δύο μας μηνύματα. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα γιατί περάσαν δύο χρόνια από τότε ότι αποφάσισε σχετικά με το να υπάρξει η τραπεζική στο Συμβούλιο και είπαμε ότι εμεί τώρα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε το υποπτικό καθήκον και την προπαρασκευή όσον αφορά τον ε, ενίο μηχανισμό ε, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Οπότε και κατά αυτόν τον τρόπο πρόκειται να βοηθήσουμε και στην ολοκλήρωση της ενιαίας ή ε, πάνω των πολλών των περισσότερων ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει ανακεφαλαιοποίηση σε εκείνες τις τράπεζες εκεί όπου ε, ανακαλύψαμε αυτές τις τρύπες στο, κεφάλαιο, αλλά επίσης τα πιο πέντε κράτη-μέλη να τηρήσουν τη δέσμευσή του τόσο ώστε να έχουν ε, μια δανειοληπτική ικανότητα ικανή, αρκετή, όπως προβλέπει το Ταμείο ε, αλλά θα πρέπει το Ταμείο επίσης να επιστρέψει και να, να, να επιστρέψει αυτά τα δάνεια και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό, αυτό ο ενιαίος κώδικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχει βοηθήσει και γι' αυτό θεωρούμε ότι τώρα θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην δημιουργία ενιαίας χρηματαγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Νούη. Και τώρα ο λόγος στις πολιτικές ομάδες και τους εκπρόσωπου του. Πρώτος ο κύριος Χάλμπα Μπιντεγκάν για το ΕΛΚ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αγαπητοί κυρία Πρόεδρε που ήρθατε σήμερα εδώ, λέει ο κύριος Μπιντεγκάιν. Ένα από τα θέματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες πολύ καλά, αλλά τους αφορούν πάρα πολύ, είναι οι πιστώσεις, τα όρια δανειοδότησης, ε, κάτι που καίει της ΜΜΕ και της οικογένειας. Είπατε ότι αύριο θα ξεκινήσει η εποπτεία για τις συστημικές τράπεζες. Αυτό όμως τι σημαίνει ότι θα αρχίσει να αρέει κεφάλαιο εποφελία αυτών των ΜΜΕ ιδίω για κάποιες χώρες όπως η Ισπανία όπου οι τράπεζες πήραν καλό βαθμό στα stress test. Δεύτερη ερώτηση κυρία Πρόεδρε. Να με υπόψη το ότι τα stress test υποχρεωτικά γιατί οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό τι σημασία έχει. Thank Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι η προσπάθεια διαφάνειας που καταβλήθηκε στα πλαίσια της περικής αξιολόγησης των τρες θα βοηθήσει τους επενδυτές να προβλέψουν την ε, χρηματοδότηση, την ε, άντληση αυτών κονδυλίων που χρειάζονται οι τράπεζες του Νότου. Πιστεύω ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη, διότι αυτό που υπάρχει στον ισολογισμό των, τραπεζών θα επιτρέψει να έχουν ταξιόγραφα οι τράπεζες που χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να περάσουν πιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές που δυσκολεύονταν έχουν πρόσβαση στην αγορά. Αυτό ήταν μια προϋπόθεση για να ξαναρχίσει η χρηματοδότηση της οικονομίας και νομίζω ότι οι επόπτες έχουν φέρει πέρα τα καθήκοντά τους ως προς αυτό. Όμως δεν είμαστε οι μόνοι παράγοντες σε αυτόν τον ε, τομέα ε, χρηματοδότησης, τροφοδοσίας της οικονομίας. Ε, η οικονομική κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά όντως συμβαίνουν. Δηλαδή θα πρέπει και οι υπόλοιποι παράγοντες να αναλαβούν δράση. Ε, σε ό,τι αφορά την, ε, τις αποκλήσεις, τα αποτελέσματα της ε, ε, σφαιρικής αξιολόγησης για τις διάφορες χώρες. Να πω ότι η όλη διαδικασία δεν αφορούσε τις χώρες, αλλά τις τράπεζες. Έχουμε μια σειρά από τράπεζε που θα πρέπει να ξαναδούν τι ελλείψει που έχουν. Υπάρχει κάποιο σχετισμό βεβαίω με την οικονομική κατάσταση τη τραπεζά του, Όταν η οικονομική κατάσταση είναι πιο ευάλωτη, η θέση των τραπεζών είναι βεβαίω πιο δύσκολη. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει κάποια, κάποια συνολική ε, ερμηνεία των δύο φαινομένων. Όμως ε, το τεστ αυτό αφορούσε τις τράπεζες και θέλαμε οι τράπεζες να βεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να προλάβουν ενδεχόμενη περαιτέρω υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Σορού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που τις αφορούν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των τεστ κόπωσης, ιδίως με το Ίδρυμα Banco di Paschi, που είχε κάποιες σοβαρές ελλείψεις. Μετά την αναγγελία των αποτελεσμάτων, ε, το 45% αύξηση του κεφαλαίου ε, έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Εκεί λοιπόν οι Ιταλοί πολίτες πρέπει να καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνουν αυτά τα τεστ κόπωσης μπορούν να πιστέψουν ε, στην αξιοπιστία, την αμεροληψία, τη δυνατότητα να δώσουν σαφείς ενδείξεις για την κατάσταση των τραπεζικών συστημάτων ε, και το πώς λειτουργεί κάθε μια τράπεζα, το κάθε ίδρυμα. Κάποιοι οικονομολόγοι διερωτώνται, και θα ήθελα εδώ μια δική σας απάντηση, πώς ε, αυτά τα τεστ κόπωσης δεν έλαβαν υπόψη και άλλους παράγοντες κινδύνου πέραν της δυνατότητας δανειοδότησης στην πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών ή την ορίμανση των ε, στοιχείων των παραγωγών προϊόντων και την ισορροπία ενεργετικου παθητικού στα στοιχεία που διαθέτει η τράπεζα. Κάποιοι έχουν ομόλογα που πολύ μεγάλης διάρκειας και αυτό βαραίνει το χαρτοφυλακιό τους ή με τα παράγωγα ε, επίσης, σε κάποιες τράπεζες υπάρχει μεγάλη δυσκολία ε, λόγω αυτών των προϊόντων. Στην ε, Μοντεπάς και τη Χένα υπάρχει κάποια ίσως μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου στο πλαίσιο, στο επίπεδο του ταμείου της τράπεζας. Επίσης, κάτι άλλο που θέλουμε να καταλάβουμε από την Ιταλική Σκοπιά είναι το εξής. Εάν δούμε τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των τραπεζών, πώς ε, επηρεάζει ότι είχε 5 δις ευρώ βοήθεια, κρατική βοήθεια το Ιταλικό κράτος προς τις τραπεζές μας ενώ είχε 240 δις ε, στήριξη το γερμανικό κράτος προς τις δικές του τράπεζες. 40 φορές παραπάνω. Είναι πρώτη φορά ε, που συμβαίνει αυτό. Ε, λήφθησαν υπόψη αυτές οι, στήρι, οι δημόσιες στηρίξεις. ελήφθη ε, υπόψη στο πόσο είναι, στέκονται καλά στα πόδια τους οι τράπεζες τις οποίες αφορούν αυτές οι βοήθειες. Ευχαριστώ. Και πάλι νομίζω ότι αφορά περισσότερο τράπεζες η όλη διαδικασία παρά χώρες, αλλά και πάλι θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αναφέρατε την Μοντε Ντεϊπάσκη. Εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτά που είπε και το Διοικητικό Συμβούλιο ε, στην ε, Ιταλία με τους Ιταλούς ελεγκτές και το τι έγινε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα. Όσοι ξέρουν ε, πολλά για, και, καλά, έχουν καλές πληροφορίες για αυτή την τράπεζα, ξέρουν ότι υπήρξε κακοδιαχείριση στο παρελθόν. Η οικονομική κατάσταση βεβαίως έπαιξε μεγάλο ρόλο στην συγκεκριμένη τράπεζα και στην κατάσταση της σήμερα. Επηρεάστηκε από το τι συμβαίνει γενικότερα στην Ιταλία, όμως Μπορώ να σας πω ότι ήταν απολύτως αμερόληπτη η όλη μας προσπάθεια με μεγάλο βαθμό διαφάνειας ως προς τη μεθοδολογία μας. Μεθοδολογία ε, ιδίω ως προς τον έλεγχο ποιότητας ε, στοιχείων του ενεργητικού που δημοσιεύτηκε. Τα κριτήρια δημοσιεύτηκαν και τα αποτελέσματα των τεστ δημοσιεύτηκαν, οπότε όντως χώρες που βρίσκονται σε δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες από άλλες βεβαίως έχουν πληγεί περισσότερο. Αυτό είναι προφανώς το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας, τέτοιου ελέγχου, αλλά προ προς τους παράγοντες κινδύνου που λάβαμε υπόψη. Λάβαμε υπόψη την πιστολιτική ικανότητα, καθώς και την δυνατότητα ε, δηλαδή με ένα τριπλό κριτήριο, για να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος εμπορίας που είναι λιγότερο διαφανής και περισσότερο αδιαφανής, ώστε να υπάρξουν απαραίτητες διορθώσεις στο επίπεδο εμπορίας και του πώς κινούνται οι τράπεζες αυτές στην αγορά. Το τεστ κόπωσης δεν μπορεί να λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες κινδύνους, είναι απλώς ε, ανέφικτο. Ιδίως για μεγάλους τραπεζικούς ομίλους σε 19 χώρες, αν σωστά θυμάμαι, και η Λιθουανία συμπεριλαμβανόταν, αλλά οι παράγοντες κινδύνου που δεν λαμβάνονται υπόψη θα ε, στο επόμενο βήμα, στη διαδικασία ε, εποπτείας, αναθεώρησης της εποπτείας, supervisory review process, ε, όπου εκεί οι συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου παραδοσιακά λαμβάνονται υπόψη σε τέτοιες διαδικασίες. Αυτό λοιπόν θα γίνει. Αυτή η διαδικασία θα λάβει υπόψη όλα τα πορίσματα των τεστ κοπόσεων, όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα, όχι μόνο τις συγκεκριμένες ελλείψεις, αλλά όλα τα διδάγματα που θα έχουμε αντλήσει από αυτήν την σφαιρική αξιολόγηση. Και από τους ειδικούς της εποπτείας θα ληφθούν υπόψη, ιδίως όσους ασχολούνται με την Ευρωζώνη, όπου υπάρχει ήδη φοβερή ενεργοποίηση και έχει ξεκινήσει ήδη σχετική διαδικασία για την ε, διαδικασία αναθεώρησης που σας λέω από τους συναδέλφους μας ε, στα ε, κράτη, τους εθνικούς επόπτες. Θα χρειαστούν όμως κάποιοι μήνες επιπλέον για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ω προ τι κρατικέ ενισχύσει υπήρξαν σίγουρα διαφορέ στην κατάσταση από τη μια χώρα στην άλλη. Εάν κάποιε τράπεζε έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να λάβουν υπόψη αυτό το δυναμικό στοιχείο στο ζυγείο τους. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία στο, ε, στο ενεργητικό των τραπεζών που εφόσον ε, φτάσουν σε μια φάση ορίμανσης πρέπει να εξαγοραστούν τελικά. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να λάβει ε, περισσότεροι θετικούς βαθμούς από τα κακά του περιουσιακά στοιχεία. Κατά την άποψή μου είχαμε ίση μεταχείριση απέναντι όλων ε, με δίκαιη ε, αξιολόγηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Αναμένουμε και τα επόμενα στάδια για να ληφθούν υπόψη όλα τα πορίσματα. Επόμενος για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Στάνισλαβ Ότζοκ. Σας ευχαριστώ Κοιτάξτε, τα σχέδια αυτά αναφέρονται σε κάποιες συγκεκριμένες ε, τράπεζες ε, και μας είπατε πως ε, προετοιμάζονται περαιτέρω μέτρα σε σχέση με όλες τις τράπεζες που συμμετέχουν ακόμα και σε αυτές οι οποίες δεν είχαν κάποιες ελλείψεις και αυτό οφείλεται ε, σε κάποια λάθη στους συλλογισμούς ή εκεί όπου διαπιστώθηκε πως ε, δεν ε, πληρείται δεν τηρείται με πλήρως η νομοθεσία. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία προγραμματίζεται. Επίσης δεν βλέπετε κάποιον κίνδυνο στην πρόταση να διαχωριστεί η επενδυτική τραπεζική από την λιανική τραπεζική. Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην πραγματική οικονομία στις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι κατά την άποψή σας ένας περαιτέρω περιορισμός της αυτονομίας των ανεξαρτήτων τραπεζών. Regarding the, capital plans. Όσον αφορά τα σχέδια για την ε, κεφαλαιακή επάρκεια πράγματι αφορούν την κάλυψη τυχών κενού, αλλά έχουμε ποιοτικέ και ποσοτικές πληροφορίες τι οποίες θα χρησιμοποιήσουμε. Πράγματι, όπως είπατε, έχουμε περαιτέρω διατάξεις, ε, συλλογικές διατάξεις ε, που προέκυψαν από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων. Κάποια από αυτά είναι λογιστικά και θα συναντήσουμε οπωσδήποτε τους ελεγκτές των ε, εταιριών για να δούμε ποιες ε, λογιστικές διατάξεις ε, θα ισχύσουν. Ένα άλλο μέρος αφορά παραδείγματος χάρη τις μη εξυπηρετούμενες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάρχουν, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι ζήτημα λογιστικού ορισμού, αλλά οπωσδήποτε αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Υπηρεσία και θα δούμε πώς θα πρέπει να υπάρξουν απαραίτητε προβλέψεις σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Τώρα για τις ποιοτικέ πληροφορίες Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, πολιτική που ακολουθείται διαδικασίες, ικανότητα να παρασχεθούν οι πληροφορίες που ζητάνε οι ρυθμιστικές αρχές εγκαίρως και με τρόπο και αυτό είναι σημαντικό. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν. Όσον αφορά τώρα τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τις τράπεζες και τον διαχωρισμό των ε, δραστηριοτήτων έχετε δει την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Ναι, κάποιες ε, αποχρώσεις, παραδείγματο χάρη, είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρατε, δημιουργία αγορών, δραστηριότητες οι οποίες στηρίζουν την χρηματοδότηση της οικονομίας πρέπει να προστατευθούν και θα πρέπει μάλλον και μάλλον θα μείνουν στο τμήμα της λιανικής τραπεζικής, όπως παραδείγματο χάρη ισχύει στο γαλλικό, στο γερμανικό δικαίο και αλλού. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να διασφαλίσουμε δηλαδή πώς θα προστατεύεται ακριβώς αυτή η δημιουργία αγοράς και βεβαίως να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι διαφορετικές εθνικές ε, νομοθεσίες ε, που προφανώς δεν ε, δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ευχαριστώ για την Άλντε Μιχαήλ Τόιρερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Νουή. Μιλήσατε για το ότι το θέμα δεν ήταν οι χώρες ε, αλλά οι τράπεζες στα stress test. Ταυτόχρονα όμως το αποτέλεσμα ε, έδειξε πως κάποιες χώρες ε, έχουν έναν υψηλότερο αριθμό τραπεζών οι οποίες θα πρέπει να συγχωνευτούν λόγω κεφαλαιακών αναγκών. Και από ό,τι φαίνεται θα οδηγήσει αυτή η συγχώνευση σε μείωση της ε, πίστης ε, σε μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Ε, συμφωνείτε με αυτή την ανησυχία μας και έχετε κάνει κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανεπιθύμητη μείωση της πίστης στην πραγματική οικονομία για να μπορέσει ακριβώς να ανακάμψει η πραγματική οικονομία στις χώρες αυτές. Και μια δεύτερη ερώτηση για τον ε, συστημικό κίνδυνο. Έπαιξε αυτό κάποιο ρόλο στα stress test, γιατί το stress test είχε εστιάσει στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πώς βλέπετε παραδείγματος χάρη την πιθανότητα αλυσιδωτών αντιδράσεων από το, τα λεγόμενα φαινόμενα ενός ε, δεύτερου γύρου στις ε, χώρες αυτές. Ε, Εάν δούμε τα στοιχεία των χωρών, πράγματι η έμφαση δίνεται στις χώρες όπου η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή ή δεν ήταν καλή. Αν και ως ένα βαθμό τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την φάση της ανάκαμψης ε, της χώρας ε, στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες. Επίσης ενθαρρυντικό είναι πως ε, οι ελληνικές τράπεζες, παραδείγματο χάρη, ε, χρησιμοποιούν το δυναμικό ισολογισμό τους. Στα σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν δεν υπάρχει σχεδόν καμία έλλειψη. Είμαστε στην αρχή της εφαρμογής των σχεδίων στην Κύπρο παραδείγματο χάρη και εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο για να υπάρξει ένα μεγαλύτερο μαξιλάρι στο δυσμενές σενάριο. Πες λοιπόν ένα μεγάλο ρόλο. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, εάν θέλουμε να αναλύσουμε την κατάσταση ανά χώρα. Αλλά ε, Κοιτάξτε, εγώ ως επόπτης ε, προτιμώ την ανάλυση ανατράπεζα. Όσον αφορά την ε, παροχή πίστοσης ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρώ πως η συνολική αξιολόγηση ήταν προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους οι τράπεζες, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία ξεκινώντας με τις μικρομεσαίες επιχείρησεις και θεωρώ πως ε, αυτό ε, τώρα σε γενικές ε, γραμμές γίνεται. Άλλα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, αυτά τα οποία είχαν γίνει με στοιχεία που είχαν ε, γίνει για την ε, εξέταση της πώληση στοιχείων που είχαν μείνει προ κρίσης. Αυτό το ξεσκαρτάρισμα των ισολογισμών μπορεί να οδηγήσει νομίζω σε μια ενίσχυση ε, των οικονομιών αν υπάρχει ζήτηση και αν υπάρχουν οπωσδήποτε επιχειρηματίες που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν. Αυτή είναι η βασική μου αξιολόγηση ότι εμείς ε, κάναμε τη δουλειά μας αλλά βεβαίως ε, και οι ε, παίκτες της οικονομίας θα πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για να υπάρξει μια νέα αφετηρία για τις οικονομίες αυτές. Ήταν προαπαιτούμενο αλλά υπάρχουν και άλλοι όροι που πρέπει να εκπληκθούν Όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο Κοιτάξτε, όταν κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο όσο η συστημική αξιολόγηση, κοιτάξτε, μεταξύ των 130 αυτών τραπεζών είναι όλες οι μεγαλύτερες, οι συστημικές, η συστημική σημασία τράπεζες της Ευρωζώνης, οπότε δεν υπάρχει νομίζω κάποια αντίφαση, κάθε άλλο, μεταξύ της ε, σταθερότητας ε, της ουσιονομικής, της ανάκαμψης, της απομάκρυνσης από τον συστημικό κίνδυνο και της ε, μακροπροληπτικής αυτής ε, δράσης που είναι η συνολική αξιολόγηση. Όλα αυτά πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Μαρίζα Ματίας για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα επανέλθω σε ένα θέμα. Θα γυρίσω σε ένα θέμα εθνικό, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά τα τεστ κοπόσεως που έγιναν στο Νόβο Banco Portugues και στην BCP με βάση ε, και όσα απάντησαν τελικά ήταν ότι δεν χρειάζονται τίποτε, ούτε κεφάλαιο ούτε ενεργετικά. Ε, ήθελα, στοιχεία του ενεργητικού δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω εσείς τι άποψη έχετε με αυτό. Και έπειτα με μια άλλη διαδικασία σε μια άλλη τράπεζα στην ε, χώρα μας, στην Πορτογαλία, την ε, BS. Εδώ δεν πρέπει ο επόπτης να προτείνει και κάποιες λύσεις όταν υπάρχουν προβλήματα στις τράπεζες. Αυτό που συνέβη στη συγκεκριμένη τράπεζα είναι ότι ε, υπήρξαν δύο παράλληλες διαδικασίες όπου όσα δεν ήταν υγιή ε, δεν ε, έμειναν στην ε, τράπεζα. Ποια είναι η άποψή σχετικά με αυτό. το κοινοτικό δίκαιο μετά από τόσες νομοθεσίες, τόσους κανονισμούς δεν απαγορεύει στις τράπεζες να έχουν και κάποια προϊόντα που δεν είναι υγιή και να τα αποκρύπτουν. Τι γίνεται λοιπόν με την εποπτεία και τις λύσεις που μπορεί να προταθούν. Ε, λυπάμαι που επιμένω στις εθνικές ε, περιπτώσεις, αλλά μας ενδιαφέρει αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα. Όντως, είναι πολύ εθνικά περιορισμένες οι ερωτήσεις σας, διότι δεν είμαστε επόπτες των τραπεζών αυτών όταν ε, δεν είμαστε μάλλον εμείς υπεύθυνοι για την υποπτία όταν προέκυψαν αυτά τα προβλήματα. Η εξυγίανσή τους έγινε βάσει του πορτογαλικού δικαίου και θα χρειαστούν ακόμη κάποιοι μήνες ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Δεν έχω πολλά να πω για όσα έγιναν στην Πορτογαλία. Έγιναν βάση των κανόνων περικρατικής βοήθειας που για την ώρα επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αλλά μέχρι εκεί μπορώ να σχολιάσω. Η ε, Μπάνκους περί του Σάντο ήταν ειδική περίπτωση. Με συγκεκριμένες δυσκολίες και δυσχέρεια να αξιολογηθεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οι άλλε πορτογαλικέ τράπεζε στο τεστ κόποση υποβλήθηκαν στην ίδια ακριβώ διαδικασία με τι υπόλοιπε, με την ίδια μεθοδολογία. Όταν υπήρχαν ε, ελλείψει κεφαλαίου, ε, αναγκάστηκαν να τι ε, καλύψουν είτε να βρουν λύσει από τον ιδιωτικό τομέα με ιδιωτικά κεφάλαια και αν όχι. Έχουμε το πρόβλημα του backstop του λεγόμενου του δημόσιου backstop και πάμε πάλι στους κανόνες περί κρατικών βοηθειών που θα ε, ε, από το 2015 με την υλοποίηση της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και την πλήρη υλοποίησή της το 2016 θα διαμορφωθούν αναλόγως. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Για τους πράσινους ο κύριος Γκίγκολτ. Καλώς μας ξανά ήρθατε κυρία Λουή. Η συζήτηση για το να ανατεθεί η εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε από τις αρχές πολλά ανοιχτά ζητήματα και αντιθέσεις. Εμείς ακολουθήσαμε αυτή την προσέγγιση μαζί με το Συμβούλιο και λόγω των συνθήκων, αλλά προείδαμε σαφώς την αρχή του διαχωρισμού μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και ο κανονισμός λέει ξεκάθαρα πως ε, αυτό πρέπει να γίνεται στο μέτρο του δυνατού. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω από εσά εάν υπήρχαν κάποια παραδείγματα όπου το Συμβούλιο της ΕΚΤ ε, άλλαξε αποφάσεις ε, του εποπτικού σκέλους. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα και τις εμπειρίας σας. Και η δεύτερη ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση. Η συνθήκη σας απαγορεύει να εξετάζεται τα ζητήματα που αφορούν τις ασφάλειες. Αλλά βεβαίως η μεγάλη τραπεζική όμιλη είναι ακριβώς αυτό, όμιλη. Πώς θα... Πώς μπορείτε λοιπόν να διαχωρίσετε αυτή την πτυχή των δραστηριοτήτων τους. Κοιτάξτε όσον αφορά τον διαχωρισμό, τις αρχές του διαχωρισμού. Εφαρμόζουμε πλήρως την αρχή αυτή, η απόφαση λήφθη από το ε, Διοικητικό Συμβούλιο για πρόσβαση στις πληροφορίες, ε, συνεργασία ή έλλειψη αυτής ε, κτλ. Όσον αφορά τώρα κάποια καθήκοντα του Εποπτικού Συμβουλίου, υπήρξε μια συζήτηση στην αρχή της συνολικής αξιολόγησης, το εάν δηλαδή αυτή ήταν κάποια προεργασία ή αν ήταν ήδη υποπτικές αποφάσεις. Κάποιοι νομικοί εξέτασαν προσεκτικά το κείμενο. Ήταν διχασμένοι. Σχεδόν μισή-μισή αυτοί που έλεγαν ε, πως ε, ήταν εποπτικοί ε, με αυτούς που έλεγαν πως ήταν προεργασία. και τελικά αποφασίστηκε πως η συνολική αυτή αξιολόγηση ήταν ε, προεργασία και άρα το Εποπτικό Συμβούλιο πάντα θα έδινε τη γνώμη του, αλλά αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο με την ε, τακτική διαδικασία. Μάλιστα. Συνέβη το εξής ε, Η μεθοδολογία βεβαίως ε, τέριαζε με αυτή τη διάκριση, αλλά ήταν σαφές στο τέλος πως οι αποφάσει, σε το αποτέλεσμα της συνολικής αυτής αξιολόγησης θα έπρεπε να γίνει με βάση μια διαδικασία ομόφωνη, χωρίς ε, αντιρρήσεις. Μάλιστα, εσείς ε, δηλαδή δεν έχετε πρόβλημα με τις παρεμβάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μήπως μπλέκουν πολύ στα πόδια σας. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, λέει η κυρία Νουή. Όσον αφορά τους ομίλους. Αυτό το εξετάζουμε με τους συναδέλφους στην ε, ΕΙΟΠΑ και ακριβώς ε, εγώ το 2010 ήμουν σε Εθνική Αρχή Επόπτης των Τραπεζών ε, πράγματι οι οποίε μπλέκονται σε ασφαλιστικές δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους που εποπτεύουν τις ασφάλειες. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν ε, ασχολείται η ΕΙΟΠΑ με αυτό το θέμα. Στο γαλλικό είναι μία η υπηρεσία, αλλά δεν αλλάζει η σχέση. Θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε αυτή τη στενή συνεργασία με την ΕΙΟΠΑ. Εγώ ήμουν και στην πρώτη συνεδρίαση, λίγες εβδομάδες ε, του πήγα στην Φραγκφούρτη και γνωρίζω πως ε, είναι αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Μάρκο Τζάνι για την EFTD. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. πρόεδρε. Ήθελα να επιστρέψω στο θέμα που έγινε και ο συνοδελφός Σόριου για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε για αυτές τις ε, αξιολογήσεις. Διότι κατά την άποψή μου ουσιαστικά δεν κοιτάξατε τους σοβαρότερους κανόνες, αλλά ουσιαστικά κοιτάξατε λίγο την επιφάνεια και εκεί την άξατε κάπως την ε, σκόνη που υπήρχε. Ήθελα λοιπόν να σχολιάσουμε την μεθοδολογία σας, WA, που χρησιμοποιήθηκε ως ε, ε, ένα μέτρο σύγκρισης. Εμείς κοιτάξαμε ένα κίνδυνο, κίνδυνο που μπορεί να παρουσιάζεται στο ισοζύγιο, κίνδυνο προ τι πιστώσει, αλλά ξεχάσαμε τελείω τι βόμβε επί τι οποίε δράζονται όχι μόνο οι ευρωπαϊκέ τράπεζε αλλά όλου του κόσμου. Τα παράγωγα δηλαδή. Τα παράγωγα είναι εργαλεία τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν βεβαίω, διότι πρόκειται για συμβάσει τόσο αδιαφανεί συχνά που είναι αδύνατο να τι κατανοήσει κανεί. Ε, ακόμα και στη διάρθρωσή του. Όμω κατά την άποψή μου, μια πραγματική ανάλυση του κινδύνου που διατρέχουν οι ευρωπαϊκέ τράπεζε θα έπρεπε να γίνει κυρίω ω προ τα παράγωγα. Ένα παράδειγμα. Εσεί θεωρείτε ότι είναι πιο επικίνδυνη μια τράπεζα. Ένα παράδειγμα τώρα, επειδή είμαι Ιταλό. Μια Ιταλική τράπεζα, όπω η Τέζα Σαν Πάολο, η οποία στο ισοζύγιο τη, στα περιουσιακά τη, έχει ω επιτοπλίστων δάνεια προ επιχειρήσει, ή μια τράπεζα όπω η Deutsche Bank, η οποία στο ισοζυγιό τη έχει παράγωγα δισεκατομμυρίων ευρώ και η έκθεση της ε, ως προς τα παράγωγα εκτιμάται στα 75.000 ε, δις ευρώ. Μια, ένας αριθμός που είναι και αδύνατο να τον εντοπίσει κανείς. Δεν τον ξέρουμε και ακριβώς. Ποια, κατά την άποψή σας, είναι πιο επικίνδυνα τις δύο τράπεζες, ποια είναι πιο εκτεθειμένη. Και υπό το φως των παρεμβάσεων, των κρατικών παρεμβάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Γερμανία δηλαδή, για να βοηθήσει την κρίση της γερμανικές τράπεζες εκταμείευσε 80 δις ε, ευρώ στην περίοδο 2008-2012. Ακριβώς γιατί οι τράπεζες ήταν πολύ εκτεθειμένες στα παράγωγα, ενώ οι Ιταλικές τράπεζες ε, ανακεφαλοποιήθηκαν από το Ιταλικό κράτος για πολύ λιγότερα δις ευρώ με ένα αριθμό πολύ χαμηλότερο από το γερμανικό. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι το πρόβλημα δεν είναι τα δανεία προς τις επιχειρήσεις, αλλά τα παράγωγα προϊόντα. Και ένα ακόμη ερώτημα ως προς το μήνυμα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με, αυτό, με αυτή την ανάλυση, με τα τεστ κόπωσης. Από τη μια θέλετε να προωθήσετε ελιγμούς όπως ε, την απόκτηση υγιών ε, περιουσιακών για να περάσουν οι ιδιωτικές τράπεζες στην ε, χρηματοδότηση, να στηρίξουν με πιστώσεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά από την άλλη, ο έλεγχο ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού, το asset quality review, δίνει ένα αντίθετο μήνυμα. Το ότι δηλαδή διακυβεύονται έτσι τα δάνεια προ τι επιχειρήσει. Ποια είναι η συνέπεια μεταξύ των δύο αυτών μηνυμάτων τελικά. Νομίζω η μεθοδολογία η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι σωστή, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κύρωση του μοντέλου γίνεται με τρόπο αρκετά συνετό. Δεν ε, γινόταν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αξιολογήσουμε αυτά που λέτε με την σφαιρική αξιολόγηση, αλλά αυτή είναι μια από τις προτεραιότητες για το 2015. Και εκεί θα αξιολογήσουμε και θα ξανακυρώσουμε τα διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στην Ευρώπη για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι σωστής ποιότητας τα, στοιχεία του περιουσιακά τους. Είναι σημαντικό αυτό για τις 18 και σύντομα 19 χώρες που ανέφερα. Δεν πιστεύω ότι τα παράγωγα είναι αναγκαστικά πιο επικίνδυνα από τις παραδοσιακές τραπεζικές ε, δραστηριότητες. Κάποιοι έχουν χάσει από τα παράγωγα, κάποιες τράπεζες, αλλά ίσως περισσότερες είναι οι τράπεζες που έχουν απολέσει πολλά λόγω της κακής ε, ανάλυσης των ε, δανείων και της κακοδιαχείρισης στα δανειά τους. Νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες κινδύνου, οι πιο παραδοσιακοί ή τα παράγωγα, πρέπει να μετρώνται με τρόπο σωστό, να είναι αντικείμενο διαχείρισης με τρόπο σωστό και να ε, αντιμετωπίζονται κίνδυνοι όπου πρέπει. Αυτό προσπαθούμε να αξιολογήσουμε όπως ε, κάναμε στη σφαιρική αξιολόγηση. Διότι τα πλέον αδιαφανή, οι πλέον αδιαφανείς κίνδυνοι στην αγορά, τα πλέον αδιαφανή παράγωγα, τα λεγόμενα επίπεδου 3, level 3 στο βιβλίο των κανόνων, είναι προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει σαφής ε, τιμή στην αγορά. Αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στην όλη διαδικασία αξιολόγησης, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά ήσυχοι με τα αποτελέσματα. Ε, νομίζω ότι σωστά ε, αυτά αντλήσαμε. Τώρα, εάν το proprietary trading ε, ή αν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι στην αγορά, εάν υπάρξει κάποιο σχετικός κανονισμός ή διαφορετικά μέτρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, θα κοιτάξουμε. Ε, να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Εδώ βεβαίως ε, το όριο είναι να μην παρέμβουμε στους ομίλους, τους μεγάλους ομίλους και τα δάνεια τους, διότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες παραγόγων στην, ε, στην κίνηση της αγοράς και περιμένουν τη βοήθεια των τραπεζών σχετικά. Εκεί τίθεται ένα όριο. Να είμαστε βέβαιοι ότι δεν εμποδίζουμε την κίνηση στην αγορά. Ευχαριστούμε ο κύριος Μονό. Κυρία Πρόεδρε, Καλησπέρα σας. Με την σταδιοδρομία σας ε, ουσιαστικά εκπροσωπείτε την τέλεια τραπεζική ε, πορεία όμως έχετε εκθέσει τους φορολογουμένους και τους καταθέτες και δεν προβλέψατε και την παγκόσμια, δημοσιονομική, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Με 25 τράπεζες στις 130 είδαμε να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και αυτό δείχνει πόσο ευάλωτο είναι το όλο μας σύστημα. Τα τεστ κοπόσεως για τις ιδιωτικές τράπεζες περιέχουν όμως και πολλά σφάλματα διότι διαπιστώνουμε ότι βασίζονται σε συστημικά σενάρια τα οποία δεν είναι δυναμικού χαρακτήρα. Τέσσερα διαφορετικά σενάρια προβλέπονται. Άμεση των ε, επιτοκίων, την αλλαγή των δανείων σε ένα κράτος μέλος και επίσης ε, την κρίση στα περιουσιακά ενός κράτους μέλους ή ενός τρίτου. Ε, αυτά τα σενάρια πιστεύω ότι είναι αρκετά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνδυασμός των σενάριων συστημικοί κίνδυνοι μπορούν τελείω να παρακονιστούν. Τρία ερωτήματα λοιπόν. Δεν πιστεύετε ότι τα συστημικά σα σενάρια, κυρία Νούγη, είναι πολύ αισιόδοξα, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν θα είναι αναγκαστικά βαθμία η σύνδεση των τεσσάρων σενάριων, αλλά μπορεί να είναι ταυτόχρονη. Τι θα γίνει επίση αν υπάρξει άλλη αντίδραση και επίσης γιατί τις ε, τράπεζες των ε, καταθέσεων, των εξοικονομήσεων τις υποβιβάζεται ενώ ε, ουσιαστικά ευνοείται τις τράπεζες των μεγάλων επενδυτών. Νομίζω ότι η πιο παλιά τράπεζα του ε, κόσμου, η Μόλτε Πάσκι Ντισιένα, είναι ενδεικτικό ότι απέτυχε στο τέσκο ποσιώσες που συγκεντρώνει τις οικονομίες των Ιταλών ε, αποταμιευτών εδώ και αιώνες. Βλέπετε ότι το κεφάλαιό της στην αγορά δεν είναι ικανοποιητικό και ουσιαστικά δεν εκπληρεί την αρχική αποστολή που θέλετε να της αναθέσετε, δηλαδή το να δανείζει μεγάλους φορείς της οικονομίας. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος τραπεζικής εποπτείας όμως. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια που αναφέρατε και τον ενδεχόμενο συνδυασμό τους, δηλαδή άμεση αύξηση των spread στα ομόλογα και ταυτόχρονα την υποβάθμιση της ελληνικής ικανότητας ειδικά στις χώρες που δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταρρυθμίσεις και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει, συνδυάζεται με έλλειψη αντιμετώπισης των αδυναμιών στα ισοζύγια των τραπεζών. Εκεί οι κίνδυνοι αυτοί όντως συνδυάζονται. Και το είπα, Α, το είπα, δεν είναι απαραίτητο ένα σενάριο που περιγράφει ένα συστημικό κίνδυνο, αλλά όσα λέγονται γύρω από αυτά τα σενάρια θεωρούν αυτούς τους κινδύνους πιο πιθανούς να προκύψουν και εκεί ε, πλήττονται περισσότερο σε μεγαλύτερο βαθμό οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν δικάνουν τα σενάρια. Αυτά τα σενάρια των αντίξεων συνθήκων έχουν ε, προταθεί από το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου της Ευρωζώνης που κοιτάζει τι γίνεται στις τράπεζες της Ευρωζώνης αλλά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, και γίνονται συζητήσεις περί των τεστ κοπόσεως και εκεί δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου SSM αλλά μόνο ρόλο παρατηρητή οπότε εγώ ακολούθησα τα τεστ κοπόσεως που προτάθηκαν αυτό μου φαίνεται ε, μάλλον ε, σωστό. Τώρα αν δυσκολεύονται περισσότερο οι εμπορικές τράπεζες και επενδυτικές από ότι οι τράπεζες των καταθέσεων δεν θα το έλεγα διότι η τράπεζα που αναφέρατε θα βρει με τους μετόχους της τα κονδύλια που χρειάζονται για να συνεχίσει, για να συνεχίσει την κλασική της, την παραδοσιακή της δραστηριότητα ως ε, τράπεζα που εξυπηρετεί την οικονομία. Εάν δούμε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην Ιταλία, διότι υπήρξε απόφαση του ε, δικαστηρίου για τις προηγούμενες κινήσεις της τράπεζας αυτής, βλέπουμε ότι ακριβώς αυτή η δράση με τα παράγωγα και η κακοδιαχείριση των παραγόγων που επακολούθησε, το εντόπισαν οι ίδιοι απόπτες της ε, τράπεζας της Ιταλίας. Οπότε νομίζω ότι αν αυτή η τράπεζα επιστρέψει λίγο στις παραδοσιακές της ε, δραστηριότητες, στήριξη των μικρομεσαίων και την ε, διατήρηση των καταθέσεων, νομίζω ότι θα γίνει και πάλι κερδοφόρα, χωρίς πρόβλημα. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε για το ΕΛΚ ο κύριος Χέις. Ε, Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε και πάλι στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα τα εξή. Αναφέρετε ότι οι, κάποιες τράπεζες, όσες έχουν ε, πρόβλημα, θα πρέπει σε 9 του να πάσουν πρόγραμμα επίλυσης των δυσκολιών τους ο οι μηχανισμός τι θα κάνει κατόπιν. Γιατί ακριβώς επειδή θέλουμε διαφάνεια θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι περιέχεται σε αυτά τα πρόγραμματα αναχρηματοδότησης. Δεύτερον, δεν θέματα που ενδιαφέρουν τη χώρα μου την Ιρλανδία γιατί έχουμε περάσει ε, ε, η βιομηχανία μας και οι τράπεζες ε, πιο πολλά θα από ότι όλες οι άλλες χώρες μαζί, αλλά η TSB, μία από τις ε, τράπεζες που πέρασε το ε, τεστ, έχει πρόβλημα κεφαλουχικό και έγινε ένα χρηματοδότηση αρκετά σημαντική του πρώτο εξάμενα. Εσείς όμως πώς βλέπετε τη συνεργασία σας με τις τράπεζες για να μπορέσετε να λύσετε κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Ας πούμε τα στεγαστικά δάνεια και το ρόλο τους στα τα δάνεια συγκεκριμένα με κειμενόμενο επιτόκιο για τη θέση τους σε σχέση με τον ισολογισμό της τράπεζας. Τι θα μπορεί να κάνει τόσο ώστε να βοηθεί η τράπεζα για να ξεπεράσει αυτές τις ε, ε, δυσκολίες ε, πρόσμα και βραχυπρόθεσμα και τι θα κάνει η Κεντρική Τράπεζα, πώς θα βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα Επίσης, πρόσφατα Πρασπιστήκατε τις θέσεις της ε, κεντρικής τράπεζας σχέση με το 20% των καταθέσεων όσον αφορά ε, τα δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Δεν θα έπρεπε ενώπιση των δυσκολιών που υπάρχουν σε αυτή τη συγκυρία να έχουμε πιο ευέλικτη ε, προσέγγιση. Αλλιώ αυτούς που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία θα τους πετάξουμε έξω από την αγορά. Αυτά τα κεφαλουχικά προγράμματα τα οποία πρόκειται να ε, μας υποβάλουν οι τράπεζες μέχρι ε, 10 ε, Νοεμβρίου πρόκειται να στείλουν το μήνυμα. Ότι δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με το κεφάλαιο και γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι με το πρόγραμμα αυτό θα καλυφθεί όσο επί το πλήστον η, τρύπα που υπάρχει. Ποιοτικέ ασφαλίσεις, μια απλή λύση και θα πρέπει οι προτινόμενες λύσει να συνάδουν προς το βαθμό κερδοφορίας τράπεζας. Δηλαδή η αγορά ε, μετοχών αντί για κουπόνια μου τότε αυτό για κάποια τράπεζα που δεν έχει πολλά κέρδη δεν είναι κάτι το λογικό. Οπότε θα δούμε. Περιμένουμε και θα δούμε. Τι θα υποβληθεί. Αλλά αυτό θέλουμε να είναι οι τράπεζες ε, ασφαλέστερες και πιο κερδοφόρες τώρα για την TSB. Ναι, και αυτή έχει πρόβλημα. Ακριβώς όπως γνωστοποιήθηκε όμως εγώ πιστεύω ότι θα εξευρεθεί λύση. Η, τώρα είναι η διοίκηση της τράπεζας. Επεξεργάζεται σχέδιο για να βρεθεί μια λύση. Τώρα αφορά αυτά τα δάνεια που είπατε, τα αστεγαστικά Εγώ ήμουν υπέρ των μέτρων που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας σας. Ζητήθηκε δηλαδή να υπάρχει loan to value. Οπότε με αυτή τη μέθοδο ήμουν εγώ υπέρ. τόσο να επανέλθει η αγορά αυτή στη χώρα σας στην ισολογική κατάσταση. Και έτσι κάποιος που θέλει να δανειστεί να μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο το οποίο θέλει. Αλλά βέβαια και στη συνέχεια να μπορεί να ρίση της υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με το δάνειο. Είδαμε με την κρίση των subprime στην Αμερική τι έγινε, πόσο φτώχινε ο κόσμος και ήταν πιο φτωχός δηλαδή αφού έπαιξε το κίνητο σε σχέση με πριν. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και έτσι να μην στριμώξουν την οικογένεια για να μπορούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Κυρία, κάνατε πραγματικά εξαιρετική δουλειά, αλλά θα ήθελα εγώ να δω λίγο σοβαρότερα το εάν επιτύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε. Είχαμε, είδαμε στην Επιτροπή μας πρόσφατα ένα πίνακα για την απομόχλευση μετά την κρίση και μάλιστα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη σύγκριση ΙΠΑ με Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι το οποίο προξενούσε εντύπωση ήταν πως πριν την κρίση η μόχλευση ήταν γύρω στο 120% του ΑΕΠ χοντρικά και στις δύο όχθες του Ατλαντικού και στις ΙΠΑ αυτό έχει μειωθεί κατά 40-50% του ΑΕΠ και στην Ευρώπη έχει μειωθεί γύρω στο 5%. Ε, αν θυμάμαι καλά. Και με βάση αυτό το συνολικό νούμερο, το οποίο δεν θα αλλάξει σοβαρά βεβαίως με βάση την ανακεφαλαιοποίηση μετά από αυτά τα οποία κάνατε, αναρωτιέμαι γιατί τα stress test αυτά ολοκληρώθηκαν επιτυχώς χωρίς ε, κάποια σοβαρά προβλήματα, αν και ε, παραδέχομαι πως υπήρχαν κάποια, ε, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια απομόχλευση. Και θα ήθελα άρα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά ένα σενάριο αποπληθωρισμού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί πως υπάρχει μια πιθανότητα 30% ε, στην Ευρωζώνη και νομίζω πως κάτι τέτοιο σημαίνει πως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν κοιτάμε το μέλλον και αναρωτιέμαι ποια θα είναι η προσέγγιση της ΕΚ όταν θα αναλάβει την υποπτία. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρθηκε ήδη κατά κάποιον τρόπο και αναφερθήκαμε στον στο ότι βασιζόμαστε υπερβολικά στα εσωτερικά μοντέλα κινδύνου και υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος ε, αν βασιστεί κανείς σε αυτά τα μοντέλα να καταλήξει σε λάθος αποτελέσματα. Βεβαίως στην έκθεσή σας 17 ε, από τις 130 τράπεζες ε, δεν εκπλήρωσαν το κριτήριο 3% της μόχλευσης της Βασιλείας 3 και μια μεγάλη χώρα από τη χώρα μου επίσης, μια μεγάλη τράπεζα και αναρωτιέμαι τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο των ε, μοντέλων και βεβαίως για να δούμε τον λόγο μόχλευσης. Ε, και τρίτον, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο τον κύριο Τόιρερ, ε, υπάρχει το βασικό ζήτημα του τι θα γίνει στην περίπτωση ε, ξεπουλήματος, εξευτελιστικές ε, τιμές που συνέβη στην κρίση και γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον ε, αν δεν λάβουμε υπόψη τέτοια σενάρια πώληση στοιχείων του ενεργητικού σε πολύ χαμηλές τιμές. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το άσχημο σενάριο προσπαθούσε ακριβώς να δει ποιες ήταν οι πιο ουσιαστικές απειλές στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Τη στιγμή ακριβώς που το κάναμε έτσι αρχές αυτού, τέλος 2013, αρχές αυτού του έτους. Τη στιγμή εκείνη το σενάριο του αποπληθωρισμού δεν ήταν βεβαίως ένα πολύτος έτσι του του λεχθέντος ε, μιλάμε για την επιθανή, τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των, του, του ποσοστού του πληθωρισμού ακόμα και κάτω από το 0. Οπότε γιατί το κακό σενάριο δεν ε, εντάξει μπορεί να μην περιέχει ακριβώς ε, ένα, την πιθανότητα πολύ αποπληθωρισμένου περιβάλλοντος, νομίζω περιέχει την δυνατότητα πολύ χαμηλού πληθωρισμού σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης. Δεν είναι ακριβώς λοιπόν αποπληθωριστικό σενάριο, αλλά έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία αυτά τα οποία θα είναι σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο. Οπωσδήποτε αρχές του 2015 θα επανεξετάσουμε τα μοντέλα όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης για να δούμε ακριβώς εάν γίνεται σωστά η εξέταση αυτών των στοιχείων. Για την ώρα βεβαίως έχουμε την σωστή βάση θα έλεγα της εξέτασης ε, της ποιότητας ε, των στοιχείων ενδεικτικών. Έχουμε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλους φακέλους ε, των δανειστών. Και εκεί πέρα ακριβώ μπορούμε να κρίνουμε την ποιότητα των χαρτοφυλακίων. Οπότε ήδη έχουμε κάνει όσα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερο θα έλεγα, περισσότερα από όσα θα έπρεπε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της εξέτασης. Για το σενάριο τώρα που αναφέρατε ως ξεπλήματος σε πολύ χαμηλές τιμές. Μπορεί να έχει παρέλθει αυτός ο χρόνος ε, για τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες. Ε, είχαμε αμέσως μετά την κρίση κάτι τέτοια φαινόμενα, αλλά για την ώρα ό,τι δεν πωλείται είναι δύσκολο να πωληθεί και θα το κρατήσουν μάλλον ε, μέχρι την λήξη του. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να ζητήσω από τους συναδέλφους να σεβαστούν ε, το χρόνο γιατί έχουμε πέντε λεπτά. Πρέπει να κάνουμε... Να περιοριστούμε λίγο. Αλέν Μασούρ, λοιπόν ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κυρία για το έργο που επιτελέσατε. Η ερώτησή μου δεν αφορά το αποτελέσματα του έργου σας, αφορά την αρχιτεκτονική, την συνολική της εποπτείας κατόπιν της ερώτησης ε, της συναδέλφου Γκίγκολ. Ε, χρειάζεται μια τέτοια ε, ενιαία εποπτεία, κάτι το οποίο το αντιλήφθη το Κοινοβούλιο πριν το Συμβούλιο. Ακριβώς ε, στα πλαίσια αυτού του πνεύματος η Κεντρική ε, Τράπεζα ε, ε, εθέσπισε αυτό τον μηχανισμό. Μετά είχαμε αυτές τις περικοπές όμως και τελικά κάνατε μια καινούργια εποπτεία η οποία είναι η υπηρεσία που εξαρτάται από την Κεντρική Τράπεζα. Άρα είναι μια περίπλοκη αρχιτεκτονική. Οπότε έχουμε εδώ τον συστημικό κίνδυνο και είπατε ότι δεν μπορείτε να πείτε κάτι διαφορετικό. Ε, και το Συμβούλιο έχει φτιάξει αυτό το σενάριο ε, της καταστροφής. Οπότε υπάρχει αυτή η υποπτική αρχή τραπεζών, υπάρχει ο ενίος μηχανισμός του, του, οποίου υγείστε και έχουμε από την άλλη μεριά τις εθνικές αρχές. Όμως δεν είναι υπερβολικά πολύπλοκο αυτό, πολύπλοκος ο μηχανισμός χωρίς να χρειάζεται με επικαλύψεις σε σχέση και με τις εθνικές αρχές. Επίσης δεν κοστίζει πάρα πολύ το να πρέπει να προσλάβετε όλους αυτούς τους εξειδικευμένους, ακριβούς συνεργάτες σε σχέση με τις τράπεζες που θα ελέγξετε και επίσης παρά την αυτονομία του μηχανισμού. Δεν υπάρχει ε, στο μέλλον ένας κίνδυνος να υπάρχει όχι σύγκρουση συμφερόντων, αλλά σύγκρουση των, των ανησυχιών, των προβληματισμών, ας πούμε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, κοιτάξτε κύριε Βουλευτά, λέει η Πρόεδρος, σε σχέση με ε, αυτού του είδους το σενάριο εμείς έχουμε λόγο και είχαμε στην ε, κατάρτιση αυτού του σενάριου αντιμετώπιση των κινδύνων και ε, ε, επειδή υπήρχε το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, δεν ήμασταν όσο δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα συνεχώς μεταβάλλονται και όσον αφορά την κατανομή των ρόλων ε, μεταξύ του, του ενιού μηχανισμού και της εποπτικής αρχής των τραπεζών. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το θέμα δεν είναι ε, το, η εφαρμοστή νομοθεσία και τα τεχνικά πρότυπα και το single rule book. Ε, εμείς εφαρμόζουμε αυτό το, το single rule book στο έργο το οποίο τελεί ο ενιαίος μηχανισμός και για την ε, τραπεζική αρχή. Επίσης δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Και επίσης συγκροτήσαμε τον ίδιο μηχανισμό με ε, δικούς μας ε, συνεργάτες και για τις πιο, πιο σημαντικές, από τις και λοιπά και έχουμε νέα επίσης από την Κεντρική Τράπεζα και οι υπόλοιποι είναι συνεργάτες των ε, εθνικών αρχών, από δηλαδή είναι κάθε τράπεζα, αλλά επίσης και κάποιες εθνικές αρχές που έχουν τράπεζες, που έχουν ε, θηγατρικές, οι οποίες ε, υπόκεινται σε, αυτόν τον, σε αυτή την υποπτία. Οπότε η συνεργασία είναι αγαστή, γιατί όλοι θέλουμε να αποδίδει αυτή η συνεργασία. Και έτσι μπορούμε να έχουμε και την πίτα χορτάτη και το σκύλο λάγερο, γιατί έχουμε τους ε, εμπειρογνώμονες, έχουμε τους συνεργάτες του δικούς μας, έχουμε τους υποπτεύοντες ε, και επίσης έτσι μπορούμε αποστασιοποιημένα να πάρουμε κάποιες ε, από την άλλη μεριά αποφάσεις για την κάθε τράπεζα, γιατί αυτή η απόσταση είναι το χαρακτηριστικό ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού. Να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτή να μειώνουν κάτι παραπάνω από του απλού τραπεζικού. Όχι, δεν είχαμε καμία ιδιαίτερη δυσκολία από αυτό. Γιατί ακριβώ, για τον ενίο μηχανισμό όλοι θεωρήσαμε ότι κάνουμε κάτι ιστορικής σημασίας. Και έχουμε συνεργάτες οι οποίοι απαρνήθηκαν πολύ υψηλότερου μισθού στον δύο τομέα για να έρθουν και να βοηθήσουν αυτό το ιστορικό έργο. Τώρα, εάν εκεί θα έχουν ε, αυτού του είδου τη θέση Σόβια, μάλλον όχι. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή. Από του Σοσιαλδημοκράτε, ο κύριο Φερνάντε. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις πρώτα-πρώτα σε σχέση με τα stress test της προηγούμενης εβδομάδας, όπως είπε ο κύριος Γιάκομ, όσον αφορά τον αποπληθωρισμό, πεστε. μας. Το Εποπτικό Συμβούλιο πρόκειται να διεξαγάγει και στο μέλλον τέτοια stress test. Αν ναι, τότε να, το, κάνετε, την εποπτεία, τον έλεγχο με πιο ρεαλιστικά σενάρια. Επίση έχουμε αυτόν τον μηχανισμό και θα έχουμε ε, ένα ξευρωπαϊσμό, εξευρωπαϊσμό, ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά, να έχουμε κάποιες τράπεζες πραγματικά ευρωπαϊκές, οπότε για να κάνουμε αυτό το βήμα σημαίνει ότι θα πρέπει να απεξεργαστούν περισσότερο το μοντέλο για τις θεατρικές που έχουμε. Κάποια φορά αποδίδει, αλλά ε, άλλες φορές ε, έχουν βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης, να έχουν κάνει ποιότερη. Να έχουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, αλλά χρειάζεται ένα πρικοδοτημένο οργανισμό επίλυση διαφορών. Ίσως κάποιο ταμείο παρακαταθήκων κοινό, ε, κάτι σχέση με το ευρώ. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Δεν έγινε στο test για τον αποπληθωρισμό. Έμεσα μόνο. Επίσης, σας θυμίζω ότι έχουμε μία σειρά από ελέγχους ο τραπεζάς που οδήγησαν σε ανακεφαλαιοποίηση που ζητήθηκε. Άρα τέτοια σφαιρική άποψη θα πρέπει να έχουμε τις κατάστασεις. Ναι, οι βοτικές αρχές χρησιμοποιούν πολύ σαν εργαλείο της δουλειάς τους τα stress test. Κάθε χρόνο. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα έχουμε τέτοιου είδους ε, τεράστια επιχείρηση με αυτού του είδους την ε, την αξιολόγηση, την ποιοτική, όπως έγινε τώρα. Θα γίνει το ίδιο δηλαδή και στα μέλλοντα stress test. Τους να το τι θα προκύψει, αφού πέσουν κεφάλια θα, θα δούμε τι θα κάνουμε και στο μέλλον. Πάντως, να δούμε τι θα γίνει για την ανασυγκρότηση και για την επίλυση των διαφορών με τη σχετική οδηγία για το ενιαίο ε, Ταμείο Επίλυση των Διαφορών. Πάντως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε οι τράπεζες να μπορούν να καλύψουν τις ελλείψεις τους με κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Εν μέρει αν όχι εν όλο. Αλλιώς θα επέμβει το Συμβούλιο με το public backstop. Γιατί το τίμημα τότε θα είναι πολύ ψηλότερο. Θα γίνει τότε βάση του δημοσίου δικαίου. Να δούμε. Θα φανεί αρχές του επομένου χρόνου. Υπάρχουν τέτοια κριτήρια τόσο περίπλοκα που δεν είμαι σίγουροι καν είναι ρεαλιστικό ότι μπορούμε να έχουμε τέτοια ανακεφαλαιοποίηση προληπτική. Οπότε θα πρέπει να πάει στην αρχή επίλυση διαφορών το 2015 η κάθε τράπεζα και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Αρχή Επίλυση Διαφόρων σκληρό, αλλά ελπίζω ότι οι τράπεζες θα καλύψουν τις ανάγκες τους από τον ιδιωτικό τομέα. κύριο Thank you, Mr. President. Uh, I have a question about uh, the development... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κίρτσος. Έχω μία ερώτηση για την πρόσφατη ανάπτυξη της σκιώδους τραπεζικής. Πολλοί αναλυτές έχουν καταλήξει το συμπέρασμα πως όσο περισσότερο ρυθμίζουμε τον τραπεζικό τομέα, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται ο σκιώδης τραπεζικός ε, τομέας ε, με τις ε, επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών ε, οχημάτων ε, και ταμείων ε, αγορών, τα επενδυτικών ταμείων αγορών που ανθούν εις βάρος του παραδοσιακού τραπεζικού τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την γνώμη σας ως ειδικού με την έννοια ότι δηλαδή για το ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τον συστημικό κίνδυνο αλλά ίσως μέσω των επιλογών μας δημιουργούμε περισσότερους συστημικούς κινδύνους. Τι θα λέγατε γι' αυτό. Ε, ε, κοιτάξτε, πράγματι όσο πιο έντονη, έντονο το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες, ε, τόσο πιο ελκυστικός φαίνεται ο σκιώτης τραπεζικός τομέας. Γι' αυτό ακριβώς στηρίζουμε τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακολουθούμε ακριβώς ε, τον ε, κίνδυνο της ε, σκιώδους τραπεζικούς, τραπεζικής. Το κοιτάμε αυτό και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, το οποίο εξηγήθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας που είναι κάποια έμεση εποπτεία της ε, σκιώδους τραπεζικής μέσω της εποπτείας των τραπεζών για τα hedge funds παραδείγματος χάρη. Ε, οι οντότητες αυτές χρησιμοποιούν τον τραπεζικό τομέα για να αποκτήσουν χρηματοδότηση ή τραπεζικές υπηρεσίες. Οπότε εμέσως, μέσω του να παρακολουθούμε στενά το τι κάνουν οι τράπεζες, μπορούμε να ελέγχουμε τον ε, κίνδυνο. Αυτό γίνεται παραδείγματος χάρη ναι, αυτό έγινε στην αρχή της κρίσης 2007-2008 με το πρόβλημα του LTCM γιατί ήμασταν ακριβώς σκληροί γιατί δεν υπήρχε τότε πρόβλημα με τα hedge funds. Ευχαριστώ κύριος Κώστας Μαυρίδης, ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νουή, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έχω τρία πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβετε, να διευκρινίσετε το σχολείο σας για το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο. Δεύτερον, θα ήθελα να φερθώ σε κάτι που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Φερνάντες σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθε. σας ρωτήσανε για τυχόν σκελετούς στους ισολογισμούς των τραπεζών και η απάντησή σας ήταν σαφής. Όχι. Ταυτόχρονα παρατήρησα πως κάποιες από τις τράπεζες που πέρασαν τα τεστ έχουν κάποια α, δάνεια μη εξυπηρετούμενα που φτάνουν το 40%. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα. Μήπως, ε, με ποιο τρόπο τα υπολογίζετε δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και κάτι άλλο. Αν δανειστώ εγώ, εγώ λεφτά εδώ στις Βρυξέλλες για το ίδιο πράγμα ε, θα με χρεώσουν 2%. Εάν ζητήσω το ίδιο δάνειο στην Κύπρο θα με χρεώσουν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι θέμα χώρας, τράπεζας θέμα ρυθμιστικού πλαισίου, κάτι άλλο. Αυτά ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για την Κύπρο όντως ε, τα stress test, ε, το άσχημο σενάριο, ξεκίνησαν ως κατάσταση ε, στο τέλος του 2013 που ήταν και ήταν ήδη αρκετά σκληρά. Σε γενικές γραμμές ε, όταν κάνουμε stress test ε, κάποιοι μας λένε πως ε, δεν ήταν καλή αυτή η χρονιά, ήταν η χειρότερη χρονιά. Εντάξει μπορεί να μην ισχύει γενικώ, αλλά πράγματι αυτό ήταν γεγονός στην Κύπρο. Τούτο λεχθέντος οι τράπεζες της Κύπρου είχαν κάποιες ελλείψεις που καλύπτονται ή έχουν ήδη καλυφθεί μέσω αύξησης ε, του μετοχικού κεφαλαίου. Ε, και αυτό είναι καλό. Αποκαθιστά την ε, εμπιστοσύνη και νομίζω ήταν καλή η συμμετοχή του στο ευρύτερο αυτό stress test που έγινε με μια ενιαία μεθοδολογία για όλες τις τράπεζες. Για το ερώτημα για τυχόν σκελετούς και ένοχα μυστικά δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν ελέγξαμε όλον τον κίνδυνο οπωσδήποτε που μπορεί να διατρέχουν τράπεζες. Αλλά αυτά τα οποία εξετάσαμε, επιστοτικό κίνδυνο, ε, κίνδυνο αγορών ε, που για τα στοιχεία εκείνα που είναι λιγότερο διαφανή και αξιολογούνται με κάποια μοντέλα Νομίζω πως ε, κατά την άποψή μου κάναμε πολύ καλή δουλειά και εγώ είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Ε, βεβαίως κάποιοι κίνδυνοι δεν εξετάστηκαν, α, νομικοί κίνδυνοι τυχόν ε, κίνδυνοι αστικής ευθύνης για κάποιες τράπεζες. Ε, δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν. Δεν τα εξετάσαμε αυτά και δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Για πράγματι τα ανοίγματα, τα μη εξυπηρετούμενα πράγματι, κάποιες τράπεζες σε κάποιες χώρες που αντιμετωπίζουν δύσκολη οικονομική κατάσταση, πράγματι είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο των ανοιγμάτων αυτών. Για να το καλύψουμε αυτό πρέπει να υπάρξει κάποια πιο συγκεκριμένη ή γενικότερη πρόβλεψη. Δεν υπάρχει κάποιο σκελετό όμως, κάποιο ένοχο ε, μυστικό. Καλύπτεται νομίζω στον ε, έλεγχο των στοιχείων ενεργητικού. Τούτ λεχθέντος βεβαίω για να είναι βιώσιμες ε, μακροπρόθεσμα οι τράπεζες πρέπει να αποκαταστήσουν την κερδοφορία τους. Αυτή είναι η ε, πρόκληση του επόμενους μήνες ε, και χρόνια. Το γεγονό ότι υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές στα επιτόκια που χρεώνουν για το ίδιο δάνειο οι τράπεζες σε διαφορετικές χώρες είναι πράγματι συνέπεια της κρίσης και της νομισματικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και νομίζω πως ε, ο έλεγχος αυτός έδωσε πολύ λεπτομερείς πληροφορίες στους επενδυτές ε, οι οποίοι θα μπορέσουν έτσι να αξιολογήσουν τα διαφορετικά επίπεδα του κινδύνου των επιτοκίων. Βεβαίως, στις χώρες οποίες χρειάζονται μεταρρυθμίσεις η επιτυχία των προγραμμάτων ε, εξαρτάται και από τις εποπτικές αρχές πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχουμε μόνο εμείς. Ευχαριστώ. Εύα Παουνόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Νούινια, ε, το σύστημα στη δική μου τη χώρα, την Βουλγαρία, και παρόλο που δεν ε, πλήγει με ιδιαίτερα από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και θεωρηθήκαμε ανθεκτικοί με την Corp Bank, ένα από τους μεγαλύτερους δανειστές στη χώρα μας, είχαμε μια τάση των καταθετών να πάρουν πίσω τις καταθέσεις τους, τη μεγαλύτερη από τη δεκαετία του 90. Θα ήθελα να είναι σαφείς και οι ερωτήσεις μου βέβαια, διότι ακριβώς ε, αυτή η τάση φυγής από τις τράπεζες οδήγησε την κυβέρνηση να οδηγήσει λόγω κινδύνου αφαιρεγκαιότητας την τράπεζα αυτή σε καθεστώς παρακολούθησης με άρση όλων της των υποχρεώσεων καθώς και την εγγύηση των καταθέσεων. Για το λόγο αυτό το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε η διαδικασία που παραβάσει κατά της Βουλγαρίας για την ε, αποτυχία της να ε, υλοποιήσει σωστά την οδηγία για την εγγύηση των καταθέσεων. Πρόσφατα, πριν από 10 ημέρες, η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Εθνικής Διαδικασίας Εποπτείας που ολοκληρώθηκε το τελευταίο τετράμενο και δείχνει ότι πρέπει να διαγράψει περίπου 2 δις ευρώ η τράπεζα αυτή σε ένα συνολικό 3,4 ενεργητικό, 3,4 δις. Με ένα πολύ μικρό ποσοστό collateral. Ε, το θέμα λοιπόν εδώ με την ποιότητα περιουσιακών στοιχείων, ε, στοιχείων του ενεργητικού στην Βουλγαρία και την ε, τοποθέτηση από τον Ιούλιο των εμπειρογνωμόνων και ε, των κυβερνητικών φορέων για την ένταξη στον SSM. Και επειδή θα ξεκινήσουν συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Βουλγαρικών Αρχών για τα απαραίτητα βήματα. Τι θα γίνει. Ε, οι βουλγαρικές αρχές δεν μας ενημέρωσαν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και τα τριμηνία αποτελέσματα του SSM δείχνει ότι κάποια κάτι μέλη μπορεί να έχουν επιφρασμένα συμφέροντα στη συμμετοχή στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και θα, δημιου... θα οργανωθούν ε, διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη ε, συμμετοχή των κρατών αυτών στον ε, μηχανισμό. Η Ευρωπαϊκή Εντική Τράπεζα λοιπόν ρωτώ, έχει γνώση των εξελίξεων στη Βουλγαρία και έχει λάβει γνώση των στοιχείων των όσων συνέβησαν. με τις νομοθετικές αλλαγές η Ευρωπαϊκή Εντική Τράπεζα πρόκειται να προσφέρει για τα τραπεζικά δάνεια την απαραίτητη νομοθετική στήριξη στη Βουλγαρία και επίση τι ενδεχομένου κινδύνου βλέπετε στην απόφαση συμμετοχή στον SSM για τη Βουλγαρία, εφόσον όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τη Τραπεζική Ένωση ούτω ή άλλω δεν έχουν εφαρμοστεί. Όντω γνωρίζουμε την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο κάποια βήματα πρέπει να γίνουν πρωτού συμμετάσχει κανείς στον ενίο αποπτικό μηχανισμό για τις χώρες που δεν έχουν και νόμισμα το ευρώ. Πρώτος είναι η υποβολή αιτήματος προς τον Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τουλάχιστον πεντάμινο προτού συμμετάσχει ένα κράτος στον ενίο αποπτικό μηχανισμό. Κατά την όσο γνωρίζω δεν έχουμε λάβει τέτοια από την βουλευτική κυβέρνηση ακόμα. Βεβαίω, ευχαρίστω και πριν λάβουμε επίσημη αίτηση να συνεργαστούμε. Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, να βοηθήσουμε τους βούλγαρου συναδέλφου εφόσον ζητήσουν κάτι τέτοιο. Για την ώρα δεν έχω λάβει γνώση τέτοιων ε, ετοιμάτων, αλλά συχνά συναντούμε τους ε, Βουλγάρους συναδέλφους και με αφορμή ε, ε και διεθνή φόρα θα δράσουμε μόλις έχουμε τις ε, κατάλληλες ε, ενδείξεις. Ευχαριστούμε κυρία Ντότση. Ήθελα να σας ρωτήσω για τις προκλήσεις συνδυασμού τον ε, τεστ κοπόσεως μαζί με τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού στη συνολική σφαιρική αξιολόγηση. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν τρεις ελλείψεις. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε ότι το EQR λαμβάνει μέρος μόνο στοιχείων, ε, ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, ειδικά επιλεγμένων για αυτή τη διαδικασία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω χάρη στον ισοζύγιο των τραπεζών μπορεί να μην ελήφθησαν υπόψη από το μέρο τη αξιολόγηση. Δεύτερον, σε ένα τέλειο κόσμο βεβαίως θα ήταν ε, σωστό να έχουν γίνει πρώτα οι, οι έλεγχοι αυτή ποιότητα στοιχείων του ενεργητικού και μετά τα τεστ κοπόσεω. Όμω τα δύο αυτά είδη τεστ έγιναν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι τα τεστ κοπόσεω δεν έλαβαν υπόψη ε, τα κατάλληλα πορίσματα όπω προέκυψαν από την έλεγχο αυτοποιότητα. Και μετά βάσει των κανόνων τη ε, ε οδηγία για τι ε, παραβιάσει στην αγορά θα υπήρχε υποχρεωτική αποκάλυψη πληροφοριών από την τράπεζα προς τους επενδυτές εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επέβαλε στις τράπεζες ε, τις ε, οδηγίες αυτές. Δεδομένων λοιπόν των τριών αυτών προβληματικών σημείων και μιας και το καθένα θα μπορούσε να έχει ε, επιρροή στην αποτελεσματικότητα της συνολικής διαδικασίας. Πώς ε, είστε βέβαιοι ότι είναι σωστά και ορθά τα αποτελέσματα της ε, συνολικής αξιολόγησης όπως έγινε, αφού δεν αξιολογήσατε τον κάθε μεμονωμένο κίνδυνο. Αισθάνεστε όντως ότι η αξιολόγηση ήταν τόσο συνολική όσο θα πρέπει να είναι σε αυτό το στάδιο. Ναι, το νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε σε κάθε τράπεζα έλεγχο του ποσοστού του ισοζυγίου που φτάνει το 60%. Τόσο πολύ ελέγξαμε. Είναι σημαντικό ποσοστό με τον έλεγχο ποιότητα στοιχείων ενεργητικού, το AQR. Επίσης, όπως σωστά είπατε, η σωστή σειρά ήταν πρώτα AQR και μετά τεστ κόπωσης. Να είναι αυτό το σημείο αφετηρία των τεστ κοπόσεω, μετά δηλαδή την ολοκλήρωση του AQR. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο. Χρειάστηκαν προσπάθειες αρκετά εφιών, αρκετών εφιών ανθρώπων στην Γενική Διεύθυνση της Δημοσιονομικής σταθερότητα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να έχουμε το μοντέλο αυτό. Αλλά ξεκινήσαμε με τα τεστ και τους αριθμούς bottom-up από τις τράπεζες, και μετά για την ε, βεβαίωση της ποιότητας, την εξακρίβωση της ποιότητας, γιατί εκεί ήταν πολλά αυτά που κάναμε, προσθέσαμε κάποια στοιχεία του AQR και μετά κάτι το οποίο το ονομάσαμε join up. Όχι απλώς μια προσθήκη δηλαδή, αλλά το ε, συνέπειες από τα όσα είχαμε ήδη εξετάσει να τα εκφράσουμε σε παραμέτρους, σε κριτήρια, κάποιες ε, προδιαγραφές για αυτά που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε συνολικά και τα τεστ κόπωσης. Νομίζουμε λοιπόν ότι κάναμε καλή δουλειά σε αυτή την προσπάθεια του Τζοϊνάπου, όπως το ονομάσαμε. Τώρα, εάν σε κάποιες τράπεζες οι επιπτώσεις του AQR ήταν σοβαρές, περισσότερα από άλλες, εκεί στις προσεχείς εβδομάδες θα μπορούσαμε να έχουμε και εσωτερική, εσωτερικό έλεγχο της λόγω τράπεζες Για να δούμε αν το 40% που δεν έχουμε ελέγξει με το AQR είναι όπως πρέπει λόγω χάρη. Θα τα μάθουμε λοιπόν αυτά αργά ή γρήγορα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για όλους τους τραπεζικούς ομίλους, για τους 30 τραπεζικούς ομίλους, μόνο για αυτές που έχουν πολύ σοβαρές να διορθώσεις να επιφέρουν ε, στο πλαίσιο του AQR. Και εκεί που υπάρχουν και απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι. Ε, έχω λοιπόν αρκετή ε, εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, έχουμε κάνει καλή δουλειά. Ήταν δύσκολη Έφτασε μια στιγμή όπου τη μεθοδολογία αυτή join up τη συζητούσαμε και δεν ήμασταν καθόλου αισιόδοξοι για το αν θα καταφέρουμε να βρούμε πραγματικά τη σωστή μέθοδο για να τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά οι συνάδελφοί μου νομίζω έκαναν υπέροχη δουλειά. Νομίζω ότι έδωσε τα σωστά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τι παραβιάσει τη αγορέ. Δεν διαφέρει πολύ από αυτό που γίνεται στον εσωτερικό έλεγχο ε, για τις τράπεζες. Υπάρχουν διαφορετικά τμήματα στι ε, σφαιρικέ αξιολογήσει. Ε, λόγω χάρη, όπω είπα, στου ελέγχου πρώτα στοιχείων του ενεργητικού βρίσκουμε κάποιε ε, ελλείψεις, λόγω χάρη στα λογιστικά, οι οποίε πρέπει να διορθωθούν ευθύ αμέσω. Η αγορά πρέπει να ενημερώνεται, διότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα να μην είναι σωστά τα λογιστικά, η λογιστική καταγραφή. Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο, πρέπει να γίνει άμεση ενημέρωση της, ε, του φορέα της αγοράς. Δεύτερο στοιχείο, η προληπτική τροποδοσία, δηλαδή η κάλυψη των προβλεπόμενων κινδύνων, ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιεί κανεί, όταν στα λογιστικά... καλύπτονται και τρέχουσε απώλειε, λίγο χάρη. Η προληπτική λοιπόν αυτή τροφοδοσία ε, επιτρέπει περισσότερο περιθώριο. Εάν είναι πολύ σημαντικά τα ποσά, πρέπει να ανακοινωθεί στους φορείς αγοράς. Αν όχι, υπάρχει περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο σκέψης από ότι στα ακρεφνώς λογιστικά. Και μετά υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο, το τεστικό στο ίδιο. Η ανάγκη να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες, ε, ενδεχόμενους τριγμούς υποβάθμισης στην οικονομική κατάσταση. Εκεί ε, δεν έχουμε ακριβώς ε, πρόβλεψη, κάποια εκτίμηση, είναι κάποια αντίξωα σενάρια που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει αν ισχύανε για κάποιο χρονικό διάστημα και εκεί ε, η διαδικασία εκτελήθηκε έτσι, ώστε όταν οι τράπεζες έλαβαν τα πρώτα αποτελέσματα, υπήρχαν σύνολα αποτελεσμάτων τα οποία ήταν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου ποιότητα στοιχείου των το EQR. Οπότε αυτά τα αφήσαμε στη στην ε, διακριτική ευκαιρία των τραπεζών. Δηλαδή, αν θεώρησαν ότι έπρεπε να ενημερώσουν τι αγορέ, το έκαναν. Δεν μπορούσαν να του πούμε να μην το κάνουν. Οι διευθυντέ των τραπεζών τα αποφασίσαν αυτά. Ε, νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και είμαι σε λογικά πλαίσια ήσυχη, διότι νομίζω ότι έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με την οδηγία για την κατάχρηση ε, των αγορών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πραγματικά εύστοχη τακτική δημόσια ακρόαση και εκτιμώ ιδιαίτερο τα όσα κάνατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην ανάληψη των νέων σας καθηκόντων αύριο. Εξαιρετική η δουλειά σας. Ευχαριστούμε και για την ε, προθυμία σας, την ειλικρίνειά σας και την παραδοχή ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θα παρακολουθούμε στενά την όλη διαδικασία και καλή σας τύχη, καλή σας τύχη στα νέα καθήκοντα της πλήρους εποπτείας. Η επόμενη τακτική μας συνάντηση στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Okay, now we next point. Ωραία, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε τη συζήτηση για τη διαδικασία στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης έχουμε την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου για τη Συλλογή Στατιστικών Πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εισηγητής είναι ο ίδιος ο Πρόεδρός σας, οπότε θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, διότι ήδη έχω παρουσιάσει τις προτινόμενες ε, τροπολογίες, την προτινόμενη τροπολογία στην πρόταση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόταση για τη διόρθωση του υπάρχοντος κανονισμού για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να καλυφθούν οι νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η ΕΚΤ μετά την δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Γνωρίζουμε ότι κατεπήγει να εγκριθεί ο κανονισμός αυτός διότι αύριο αναλαμβάνονται αυτές οι νέε αρμοδιότητες ακριβώ. Το σχέδιο πράξης επιτρέπει να αξιοποιούνται από την ΕΚΤ οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες ανάλογες με αυτές που έχουν οι εθνικές τράπεζες στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας που πρέπει να ασκεί. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί να αποστέλει εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και στις εθνικές αρχές που ασχολούνται με την εθνική εποπτεία στα πλαίσια της σταθεροποίησης του ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος ε, και του ενιαίου μηχανισμού. Ε, το σχέδιο εκθεσή μου μιλά για την. δύο τροπολογίες. Η νέα περιορίζει τις νέε αρμοδιότητες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Και η δεύτερη προβλέπει απαιτήσει για τι αρχέ που λαμβάνουν τι εμπιστευτικέ στατιστικέ αυτέ πληροφορίε, να λαμβάνουν δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιώνονται για την προστασία αυτών των πληροφοριών. Αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 21. Έχει διορθωθεί ώστε να καλύπτει καλύτερα τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να φροντίζουν τα εμπιστευτικά στοιχεία που αποστέλλονται στο ε, σύστημα είναι ε, προστατευμένα. Έχουμε λάβει 19 τροπολογίες, θα κριθούν βάσει του ε, εάν θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο της διαβούλευσης, όχι μόνο στη συγκεκριμένη αρμοδιότητα επικαιροποίηση του κανονισμού εν ώψη του, του κανονισμού για τον ε, ε, ενίο υποπτικό μηχανισμό ή να τον περιορίσουμε. Να περιορίσουμε το πεδίο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθεί τώρα η Επιτροπή μας. Ε, πολύ σύντομα να σχολιάσω κάποιες από τις τροπολογίες. Ούτως ή άλλως έχουμε και τις εξηγήσεις των ε, όσων πρότειναν τις ε, τροπολογίες. Για τις τροπολογίες του κ. Μπάλτ 5, 6 και 8 συγκεκριμένα για την πέμπτη, για τη συμπερίληψη της σχετικής ε, διάταξης, για, την, ε, για τις λογιστικές προδιαγραφές την ε, νομοθεσία της Ένωσης, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη στην αγορά και το απαραίτητο πεδίο για τη συλλογή δεδομένων. Εδώ θα θέλετε να μου το εξηγήσετε πώς το εννοείτε αυτό με, το, με την κάλυψη της αγοράς και επίσης για την τροπολογία 6 τι εννοείτε με το reporting channel, το διάβλο ενημέρωσης. Πώς ακριβώς το εννοείτε όσο για την τροπολογία 8. Συμφωνώ απολύτως με την πρότασή σας οπότε νομίζω χρήσιμο θα είναι να υπάρχει μνήα της αρχής τη αναλογικότητας. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του κυρίου Φερνάντες. Αυτές έχουν περισσότερο στόχο να διευρύνουν το πεδίο της διαβούλευσης, της όλης διαβούλευσης, Αυτό λοιπόν είναι εναπόκειται στην δική μας απόφαση να θα ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση όχι. Αν ναι, εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι να πάμε προ αυτή την κατεύθυνση Θα κάνω και εγώ τα ανάλογα σχόλιά μου, δηλαδή για την τροπολογία 4. Η δημοσιοποίηση εξαιρέσεων ε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τους ε, υπεύθυνους των εκθέσεων. Η ανάγκη εκπαίδευσης και εργαστηρίων ε, στην, στην ε, ναι, δεν ξέρω αν είναι κάτι που μπορούμε να αποδεχθούμε, αλλά ένα άλλο μέρος της ΝΕΣ, την τροπολογία 10, είναι κάπως μεγάλη υποχρέωση αυτή, το raw data, αλλά μπορώ να το αποδεχτώ. Στην τροπολογία 11 η δυνατότητα να γίνουν συγκριτικές στατιστικές αναλύσεις νομίζω ότι ξυπακούεται στις αρμοδιότητες της ΕΚΤ, δεν ξέρω αν υπάρχει ανάγκη τέτοιας τροπολογίας. Θα ήμουν πιο συνετός με την τροπολογία 12 για την ε, δημοσιοποίηση των ε, εκθέσεων παραβιάσεων. Είναι νομίζω ευαίσθητο στοιχείο αυτό για να δημοσιοποιείται έτσι απλά. Για τις 13 και 14 κατά την άποψή μου δεν είναι απαραίτητες διότι η κακοδιαχείριση παραποίηση στοιχείων ούτω ή άλλω καλύπτεται από τον ορισμό των ε, συλλεγόμενων στοιχείων, κατά την άποψή μου. Περισσότερο νόημα θα είχε να ε, ε, ενημερωθεί το επίπεδο των προστήμων όπω προτείνουν οι τροπολογίε 15, 16 και 17 καλύτερα. Ενώ από την άλλη νομίζω ότι είναι εκτό πεδίου απονομική άποψη να προβλεφθεί ένα αυτόματο μηχανισμό επικαιροποίηση όπως ε, υπονοεί η τροπολογία 20. Νομίζω η τροπολογία 18 μπορεί να γίνει αποδεκτή, ενώ η 19 δεν νομίζω από νομικής πλευράς να είναι εδώ το σημείο που θα πρέπει να προβλέψουμε μια τέτοια προπόθεση, μια τέτοια απέτηση. Αυτά είναι τα σχόλιά μου για τις τροπολογίες. Είμαι βεβαίως ανοιχτός να ακούσω τα σχόλιά σας και να ε, προσπαθήσω να συνδυάσω τις διάφορες απόψεις με συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ καλή σας δουλειά. Θα είμαι σύντομος. Εγώ θεωρώ πως οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. Γι' αυτό και υποστηρίζω ρητός τις τροπολογίες του εισηγητή, όπως ακριβώς τις ε, παρουσιάσατε τώρα. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω τις ανησυχίες μου, τις επιφυλάξεις μου για το πόσο ε, ευρεία μπορεί να είναι αυτή η συλλογή δεδομένων της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Ε, ανέφερα ήδη και το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε πως ε, είναι ουσιαστικό ζήτημα εδώ η αναλογικότητα. Κατά την άποψή μου πρέπει να διασφαλίσουμε πως η υποχρέωση αυτή πληροφόρησης ειδικά όσον αφορά τις, ε, μικρο, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, ε, να μην ε, οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των αναφορών που είναι υποχρεωμένο κανείς να υποβάλει στις αρχές εξού και οι τροπολογίες 5 και 6. Θα πρέπει να παραμείνουμε στις γνωστές συνήθεις αναφορές. Όσον αφορά αυτά τα οποία αποφασίσαμε ήδη στην τομεακή οδηγία, δεν θα πρέπει να τα ανατρέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος, κατά την άποψή μου, είμαι κατά της αύξησης των ε, κυρώσεων ε, όχι βεβαίως υπέρ του μηδέν που λένε οι συνάδελφοι, απλά νομίζω καλό είναι να υπάρχει μια διαβάθμιση. Θα έλεγα. Αυτές ήταν οι δικές μου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω για το ECR. Ναι, παρακαλώ. Η κόρα. Ναι, και Ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα στις παρατηρήσεις του Προέδρου. Όπως είπα και στην ανταλλαγή απόψεων, εγώ θεωρώ πως θα πρέπει όλες οι εποπτικές αρχές ε, να χρησιμοποιούν τα καλύτερα ε, διαθέσιμα δεδομένα και έτσι θα έχουμε και καλύτερη πρακτική. Επίσης συμφωνώ με τον Πρόεδρο στο να έχουμε μια, ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να περιοριστούμε εδώ στο στον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό. Έχω κάτι το οποίο μπορεί να σένεται λεπτομέρεια και έτσι σχολαστικότητα. Αλλά εγώ θα ζητούσα η τροπολογία υπαριθμών 19 του κυρίου Φερνάντες να συμφωνεί με οτιδήποτε αποφασίσουμε στην επόμενη έκθεση. Δεν θέλω τα πρόστιμα να διαφέρουν από τη μία έκθεση στην άλλη. Να το συζητήσουμε στην επόμενη έκθεση και να είναι τα ίδια και εδώ. Ευχαριστώ. Πράγματι, μάλιστα, άλντε τώρα. Η κυρία Κόρα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ σύντομη. Σε γενικές γραμμές βεβαίως οι προτεραιότητες είναι να διασφαλίσουμε την ε, εμπιστευτικότητα και την αναλογικότητα και να μην επιβάλλουμε υπερβολικό βάρος ε, στις επιχειρήσεις. Να υπάρχει δηλαδή μια λογική προσέγγιση όσον αφορά τις κυρώσεις. Για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών συμφωνούμε πως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα στηρίξουμε τις τροπολογίες εκείνες που θα ενισχύσουν την ε, εμπιστευτικότητα των δεδομένων που θα δοθούν. Για την αναλογικότητα τώρα είναι επίσης σημαντικό να ασφαλίσουμε πως οι νέες απαιτήσει ε, θα είναι αναλογικές και να μην υπάρχει υπερβολικό βάρος ε, στις επιχειρήσεις αυτές. Και τέτοιες τροπολογίες θα στηρίξουμε λοιπόν για τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις για τη μη παροχή ακριβών δεδομένων πρέπει να είναι σαφείς, απλές αποτελεσματικές και όχι υπερβολικές. Οπότε η μεγάλη αύξηση των κυρώσεων μας φαίνεται κάπως υπερβολική και το να δημιουργήσουμε ένα διαφοροποιημένο σύστημα κυρώσεων είναι κάτι το οποίο περιπλέκει τα πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν βλέπουμε το, το λόγο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ δεν βλέπω πουθενά την Μαρίζα Ματίας ή κανέναν από την ΚΟΕ. Α, Σβέν. Όχι, δεν υπάρχουν σχόλια από τους πράσινους. Γιώνας, θέλεις το λόγο. Μάλιστα ήταν σύντομη συζήτηση αλλά σαφής. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τις παρεμβάσεις. για την ε, ενίσχυση της εμπιστευτικότητας και βεβαίως ε, συμφωνώ πλήρως με αυτό το είπε η ΚΕΙ ότι πρέπει να δούμε το θέμα των κυρώσεων να είναι ίδιο με την άλλη έκθεση για την ε, αύξηση, την αυστηροποίηση των κυρώσεων βλέπω πως υπάρχει κάποια θέση δύο-τριών ομάδων και βλέπω μία τάση να προσπαθήσουμε να μην διαβρύνουμε πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογή. Αντιλαμβάνομαι επίση αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Μπάλσης. Ε, Διαμφιβολία μου τώρα για την τροπολογία 5 μπορούμε να το δούμε. Για την 6 μπορούμε να το δούμε ατομικά νομίζω, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια συνένεση για τη γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και κάποιον συμβιβασμό στον κατάλογο ψηφοφοριών. Αυτά αρκετά νομίζω με αυτή την έκθεση μα με συγχωρείτε, η ψηφοφορία στις 11 Νοεμβρίου μαζί με την ψηφοφορία της άλλης έκθεσης ε, που πάει μαζί η εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δηλαδή για επιβολή κυρώσεων και δίνω τον λόγο στην Κέι Σουίνμπορν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις τροπολογίες. 25 είναι μόνο. Άρα δεν θα είναι και τόσο δύσκολο τώρα να τις συζητήσω όλες γιατί στα περισσότερα συμφωνούμε οπότε τελικά συμφωνώ σχεδόν με όλες αυτές που προτείνατε. Έχουμε όμως λίγες εξαιρέξεις. Εκεί πάντως που υπάρχουν περισσότερες διαφωνίες είναι η 15 μέχρι τη 18. Εκεί που λέει <clears throat> την δημοσιοποίηση των κυρώσεων. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να μην γίνει η δημοσίευση αυτών ε, κατ' επιλογή. Είπαμε, ε, πολλοί έχουν έρθει και μου έχουν πει και μου έχουν γράψει ότι κάνω λάθος, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι υπάρχει συνένεση, ότι δηλαδή η αρχική πρόταση μας οδηγεί σε ένα παράδειγμα επίπεδο ε, απορρίτου υπέρ της ΕΚΤ. Απαντός θα πρέπει να δούμε κατά πόσον, όχι ας μη συμφωνεί η ΕΚΤ, εμείς εδώ να τα βρούμε. Επίσης, ξέρω, επειδή έχω δουλέψει και στον ε, κανονισμό για την καταχρηστική λειτουργία στην αγορά θα πρέπει να υπάρχει μια επιλογή όσον αφορά κάποιες ε, παρατάσεις, όποτε υπάρχει κάποια διατάραξη της αγοράς, οπότε και εγώ συμφωνώ για το ότι χρειάζεται να υπάρχει κάποιο είδου ε, ε, χρονισμός επιβράδυνσης και θα πρέπει να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορεί να αναβάλει η Κεντρική Τράπεζα αυτές τις κυρώσεις ή κατά πόσον μπορεί να τις επιβάλλει γρηγορότερα. Να το δούμε αυτό τις επόμενες μια-δυο μέρες, εάν μπορέσετε, στείλτε μου τη γνώμη σας. Α, τώρα, τώρα, μου τελειώσει η συνεδρίαση για να δούμε κατά πόσον, τι λέτε. Ε, δηλαδή τα δύο χρόνια είναι πολύ, είναι λίγο, να προτείνει κάτι άλλο, μικρότερο, ε, πιο μακροχρόνιο. Πάντως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και την περίπτωση της αναβολής της δημοσίευσης, πάλι θα πρέπει να υπάρξει ε, μία συζήτηση εδώ στο Προεδρείο της Επιτροπής μας για να δούμε εμπιστευτικά τι έχει γίνει και γιατί υπάρχει η αναβολή της δημοσίευσης. Και οπότε θα πρέπει από την μηδενική καθυστέρηση πάμε μέχρι τα πέντε χρόνια. Οπότε και εγώ θέλω να δω ε, εσείς τι πιστεύετε πόσο μεγάλη αναβολή θα πρέπει να υπάρχει Τι λένε οι πολιτικές ομάδες. Συνδεσμός θα μπορούσε να βρεθεί εάν σήμερα συμφωνείτε ιδάλλως στις επόμενες μία-δύο μέρες και να κάνουμε ανταλλαγή απόψε και τελικά καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική περίοδο να βολεστώ όσον αφορά τις τεχνικές ε, ε, ε, τροπολογίες κύριε Γκίγκολτ είπε κάτι σε σχέση με την ευθυγράμμιση με τον ενίο μηχανισμό SSM και ε, κατάλαβα σωστά, νομίζω ότι συμφωνούμε. Και όσον αφορά την διαφάνεια, προτείνει εδώ και όσον μια, ε, μια διαδικασία που συμφωνώ, διότι νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοια διαφάνεια. Γιατί θα κάνουμε σε σχέση με αυτή την εφαρμοστεία διαδικασία όσον αφορά ε, την αναβολή και δεν θα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα, να μην γίνεται κατά περίπτωση ε, ο, ο χειρισμός. Κανόνες προβλέψιμη και με διαφάνεια. Για όλους. Και ίση μεταχείριση για όλους και απουσία δυσμένους διάκρισης. Επομένως είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει ένα πλαίσιο και έτσι να μπορεί να ενεργήσει ε, με τρόπο που να θεωρείται άψογος και να υπάρχει και μια διαδικασία προσφυγής ε, η οποία να μην αναθεωρηθεί την επαύριο. Επίσης, θα δούμε τι γίνεται με τις δημοσιεύσεις, να μην υπάρχει μεταξύ της τροπολογίας 6 της δικής μου και σχέση Κίγκολτ υπαριθμών 23. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ε, το ότι και οι δύο φορούν το ίδιο πράγμα. Να κάτσουμε και να δούμε όμως την διατύπωση. Παρακαλώ ας βοηθήσει για τη διατύπωση η γραμματεία. Και να δούμε τι διατύπωση μπορεί να περάσει, αλλά και ταυτόχρονα που να περνάει το μήνυμα το οποίο θέλουμε. Στεγανή διατύπωση όμως να βρούμε. Αποδεκτή όλους τώρα να δούμε μία-μία τροπολογίε εκεί που περισσότερο δυσκολεύτηκα αφορούσε τι τροπολογίες 19 και του κυρίου Φερνάντε. Εδώ υπάρχει παραπομπή στην προηγούμενη έκθεση και να δούμε τι γίνεται, πού πάνε τα έσοδα από τις χρηματικές ποινές. Πέστε μου. Εγώ αρχικά θεώρησα ότι θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρηματοδοτήσει τις έρευνες. Τα νομικά έξοδα στην άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων, αυτό θα γινόταν σε κάθε περίπτωση ε, σε εθνικό επίπεδο. Να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με το πώς δαπανώνται τα έσοδα. Είναι σημαντικό. Έτσι αυτό να μην είναι παράγον που γεννά κεφάλαια και έσοδα για την ε, Κεντρική Τράπεζα. Οπότε παρακαλώ να μου εξηγήσει ο κύριος Φερνάντες πώς το είδε ακριβώς και αν συμφωνεί εκείνο, αλλά και οι άλλοι για το κατά πόσο πρέπει αυτά τα χρήματα να πηγαίνουμε στην Κεντρική Τράπεζα. Πού να πάνε, να πάνε στο κατευθείαν στον κοινωνικό προπολογισμό, να πάνε στο Ταμείο Επίλυση Διαφόρων. Συμφωνώ με την 25 και με την 13 τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά αυτέ τι κυρώσει. Και αυτό το διαπιστώσαμε ότι ισχύει για πολλά διασυνοριακά διεθνή σκάνδαλα. Το διεθνέ έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα. Οπότε θα πρέπει οι πολιτικέ αρχέ να συνεργάζονται για να υπάρχει ένα σύστημα στεγανό για την εφαρμογή των χρηματικών ποινών. Τώρα έχουμε το 11. 11 για αποφυγή δυσμενών διακρίσεων είναι σημαντικό να δούμε το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση στο σύστημα και έχουμε στον μηχανισμό ε, κάποιες ε, διατάξεις που εδώ πέρα συντρέχουν Ό,τι μου λένε όπως έχει τώρα το κείμενο δεν συνάδει 100% με τον ενίο μηχανισμό SSM. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την νομική βάση, κατά πόσο όλα αυτά είναι σύμβατα με τον SSM και τι μπορούμε να κάνουμε για να το διορθώσουμε αυτό. Δεκατέσσερα, Φέρμπερ. Εδώ προβληματίζομαι κάπως. Εγώ κατάλαβα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει την αρμοδιότητα που είχε προηγουμένω ε, η Τραπεζική Ένωση. Να δούμε. Μήπω οι εθνικέ αρχέ είναι τελικά αρμόδιε. Να δούμε τι λέει το κείμενο για την Τραπεζική Ένωση. Ποιο αποφασίζει ότι πρέπει κύρωση και ποιο εφαρμόζει την απόφαση. Βέβαια, υπάρχει νομική παράδοση, νομική ένωση και λέμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η Εθνική Αρχή της κυρώσεις και εδώ πέρα σας παραμείνουμε στην τροπολίνη παριθμών 3 που νομίζω ότι θα άρεσε και θα καλύψει τον κύριο Φέρμπερ για να βρούμε την ε, ισορροπία μεταξύ των Εθνικής Αρχής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζω ότι αφού σας ακούσω θα καταλήξουμε σε συμβασμό, έχω να προτείνω εγώ τρεις συμβασμούς, που νομίζω θα σας βρουν σύμφωνους και νομίζω ότι θα ψηφίσουμε όπως είχαμε πει την επόμενη τρίτη αυτή την έκθεση. Νομίζω κανείς θέλει να ε, αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της Τραπεζικής Ένωσης. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το κείμενο, αν όχι τότε ζητάω πολλά. Και σε ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα δώσουμε το, ρωτο λόγο στον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ και την ΚΕΙ για τη δουλειά που έκανε. Αν δει κανείς τις τροπολογίες επικεντρωνόμαστε σε τρία θέματα ποιο είναι το σωστό μέτρο διαφάνειας, ειδικά όσον αφορά την δημοσίευση των κυρώσεων. Δεύτερον, τι θα γίνει με την παραγραφή, πότε ξεκινάνε οι προθεσμίες, ποια είναι τα κριτήρια, αν μπορεί να διακοπεί και το τρίτο θέμα είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Και βεβαίως έχουμε κάνει εδώ πέρα τροπολόλα Όσον αφορά την διαφάνεια, επί της αρχής νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε διαφάνεια, αλλά ήδη είπα πως ε, διπλή τιμωρία και από την αγορά και από το κράτος, δηλαδή και από τις υποπτικές αρχές και από την αγορά, ε, λόγω της ε, πολύ γρήγορης δημοσιοποίησης θα πρέπει να αποφευχθεί νομίζω μία τιμωρία αρκεί. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε κάπως συγκρατημένοι. Εγώ έχω υποβάλει μια τροπολογία ε, η οποία λέει πως θα πρέπει να δημοσιεύεται η ποινή μόνο όταν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα. Το βρίσκω λογικό. Γιατί η εμπειρία το παρελθόν δείχνει πως ε, πάντα προσέχουν στα δικαστήρια οι ενδιαφερόμενοι και προσφέρουν και την ουσία και τα θέματα αρμοδιότητας κτλ και βεβαίως όσο είναι στα δικαστήρια δεν ε, ισχύει η ποινή, οπότε δεν χρειάζεται να δημοσιευτεί όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής. Νομίζω πως ε, πράγματι βλέπουμε πως ε, περνάει πολύ καιρό για να ανακαλυφθούν ε, ε, κάποια διοικητικά λάθη, οπότε δεν θα πρέπει να περνάει να, πάρα πολύ γρήγορα η προθεσμία της ε, παραγραφής τώρα. Το, εάν θα είναι η αρμοδιότητα της ΕΚΤ ή όχι... Κοιτάξτε, Το θέμα είναι βεβαίως και πού θα μπορεί κανείς να προσφέρει εκεί στα δικαστήρια. Έτσι. Και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σε όσοι ασχοληθούν με αυτό. Και πραγματικά και η χαρά σκουράγιο σου που ασχολείσαι με ένα τέτοιο θέμα που είναι και τη Ευρωζώνη. Αλλά βεβαίω. Εντάξει, θα πρέπει να ε, υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά να επιβάλλουν ποινές μπορούν, νομίζω, μόνο οι εθνικές αρχές, έτσι, ποιος έχει την ε, αρμοδιότητα ε, και την αρμοδιότητα ε, και την νομική βεβαίως έτσι. Δεν τώρα θα μπω εγώ στο, στη λογική αυτή του πόσα χρόνια χρειάζονται ούτε στην αριθμητική αυτή λογική. Εγώ θεωρώ πως η, δική μου βεβαίως η τροπολογία είναι η σωστότερη, κατανοητό, αλλά εντάξει θα το δείξουν αυτό οι ψηφοφορίες. Ε, νομίζω πως αναφέρθηκα στα ουσιαστικότερα σημεία. Βεβαίως ε, είμαστε και στη διάθεση της εισηγήτριας για διμερείς ε, συνομιλίες. Ευχαριστώ. Ο Κώστας Μαυρίδης από τους Σοσιαλδημοκράτες. Σκιώδης ναι. Όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή, δύο σύντομα σχόλια. Για την τροπολογία 9 συμφωνούμε όλοι πως η διαφάνεια πρέπει να είναι προτεραιότητα, αλλά βεβαίως υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις και συμφωνούμε πως η αιτιολόγηση που υπάρχει εδώ είναι επαρκής, αλλά πρέπει να επιβάλλουμε την ίση μεταχείριση για όλες τις τράπεζες ανεξαρτήτως μεγέθους. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής. Η τροπολογία 11 για το επίμαχο κείμενο, για το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα προωθήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό. Αυτό το οποίο προτείνω είναι να υποβάλω μια προφορική τροπολογία που θα χωρίζει αυτό το κομμάτι του κειμένου σε διαφορετική, σε χωριστή πρόταση από το άρθρο 8. όσον αφορά την τροπολογία 6. Εάν έπρεπε να επιλέξω, η διατύπωση για την ε, έναρξη διαδικασίας υπαραβάση παραβάση ε, είναι αυτή την οποία θα προτιμούσα και ο λόγος είναι ο εξής περιορίζει την οποιαδήποτε υποκειμενικότητα σε σύγκριση με την διατύπωση που είδα σε κάποιες άλλες ε, τροπολογίες δεν ξέρω αν είμαι σαφής μπορούμε να το συζητήσουμε ναι ωραία αυτά σας ευχαριστώ Κόρα από την Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα το εύλογο χρονικό διάστημα για τη δημοσιοποίηση των κυρώσεων, ώστε να υπάρχει σαφήνεια για την αγορά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι αντικείμενο εποπτεία από την ΕΚΤ. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη απόφαση την ΕΚΤ για τι κυρώσει και τα πρόστιμα. Θα πρέπει οι διαδικασίε αυτέ να είναι κατανοητέ, εύληπτε, διαφανεί και να ολοκληρώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσω την ε, Σκιώδη λοιπόν για τη δουλειά της ως προς όλα αυτά τα θέματα. Για τη δημοσιοποίηση λοιπόν των ε, κυρώσεων ως γενικό κανόνα νομίζουμε η ΕΚ θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων. Όμως η ΕΚ θα πρέπει να έχει την διακριτική ευκαιρία να μην δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις ε, εντός προϊόντος συγκεκριμένων προθεσμιών, εφόσον δεν είναι τελική απόφαση και δεν έχουν οι δυνατότητε ε, άσκηση έψη. Για τι περιόδου κάλυψη των προστήμων και τη πληρωμή του, θα πρέπει να ε, δώσει περισσότερο περιθώριο η ΕΚΤ από ό,τι έχει προταθεί αλλά τα καθημερινά η διάκριση των προστήμων σε καθημερινά και με καθημερινά δεν είναι μια λογική διάκριση. Ως προς τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων θα θέλαμε να παραμένουμε στα παραδοσιακά πλαίσια του περιορισμού για τις Αθήνα προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή οι κυρώσεις και οι αποφάσεις για αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή πέντε χρόνια μετά την παραβίαση, όπω προτείνει και η ΕΚΤ. Η διακοπή αυτού του χρονικού πλαισίου θα πρέπει να δικαιολογείται εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Όπως η πρόταση που κάνει η ΕΚΤ. Η πενταετής ε, διακοπή που προτείνει η ΕΚΤ. Κατά τα άλλα, μπορούμε να δεχτούμε τις τροπολογίες που βάλει ο κ. Φαμπέ και ο κ. Μπάλτς. Αυτά. Thank Ευχαριστούμε. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ. Μόλις έφτασα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν άκουσα το ε, υπόλοιπο της συζήτηση που έγινε. Δεν είμαι σχεδόν εισηγήτρια για την έκθεση αυτή από την ΚΟΕ. Ε, ο συνάδελφος Βιέγκας δεν μπορούσε να είναι εδώ, απλώς να κάνω κάποια σχόλια γενικότερο χαρακτήρα ό,τι έχει να κάνει με την προσέγγιση μιας τέτοιας έκθεσης της Γνωρίζω ότι πολλές φορές είμαστε πολύ ε, αστεροί σε σχέση με το τι δραστηριότητες έχουμε εδώ υπόψη μας, όμως δεν πρέπει να πάψουμε τη σοβαρή ε, αξιολόγηση της πολιτικής που προτείνεται και υλοποιείται από την ΕΚΤ. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που με ανησυχούν αρκετά. Πρώτα απ' όλα ότι αν δεν γίνει αυτή η σοβαρή αξιολόγηση της νομισματικής μας πολιτικής και της αποτελεσματικότητάς της και σε ε, συνδυασμό με άλλες πολιτικές που υλοποιούμε, τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να είναι πάντα τα ίδια. Ακόμη και αν ανακοινώνονται θετικά αποτελέσματα, η νομισματική μας πολιτική ως τώρα ήταν καταστροφική. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πρέπει να υπάρχει μια έπρεπε να υπάρξει μια τεράστια τροφοδοσία ε, κεφαλαίων προς τις τράπεζες, φτηνό χρήμα που έφτανε στις τράπεζες αλλά όχι στην πραγματική οικονομία, ακριβώς διότι η ζήτηση και η προσφορά δεν είχαν ακόμη εξισορροπηθεί. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη ζήτηση ακόμη και εάν συνεχίσουμε την νομισματική μας πολιτική που είναι τόσο επεκτατική αλλά δεν επιτρέπει το χρήμα να φτάνει στην πραγματική οικονομία, τότε οι τράπεζες θα μένουν χωρίς χρήμα και κάτι θα πρέπει να κάνουν. Τι είναι αυτό που θα κάνουν. Αυτό που πάντοτε ανέκαθεν έκαναν. Κερδοσκοπία πολιτική κερδοσκοπική. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά είναι τελείως αδύνατο να διαχωριστούν. Νομίζω ότι σε μια έκθεση για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ πρέπει ακριβώς να κοιτάζουμε, να υποβάλουμε συγκεκριμένε χειροπιαστές προτάσεις, ως προς την ανάγκη λόγω χάρη να υπάρχει ένα πόλη σε μίξη, μια ανάμιξη, ένα συνδυασμό πολιτικών, ώστε να ξεφύγουμε από την τροχιά που έχουμε ακολουθήσει ως τώρα και να περάσουμε σε μια θετική χάραξη πολιτικής. Μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη αποτυχία. Καμία επίτευξη των στόχων προτείνονται. Πρόεδρος. Νομίζω είσαστε σε λάθος σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δεν μιλάμε για την ετήσια έκθεση τη Κεντρική Τράπεζα. Πω, πω, με συγχωρείτε. Μιλούσα για το επόμενο. Ε, έκανα ήδη την παρέμβασή μου. Μόλι είχα φτάσει, δεν με ειδοποίησε κανεί γιατί μιλάμε. Εντάξει, έκανα λοιπόν την παρέμβασή μου για την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα έχω τίποτα να πω στο επόμενο σημείο. Για τι κυρώσει δεν έχω να σχολιάσω. Με συγχωρείτε. Εντάξει, το σημειώνουμε πάντως, σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας. Επόμενος ομιλητής, θέλετε να πείτε κάτι για το σημείο αυτό. Όχι, ωραία. Περνάμε στον Σβέν. Σβέν Γκίγκολτ. Ανακουφισμένος αισθάνομαι, γιατί νόμιζα ότι θα αρχίσουμε μια εφόλης της ύλη κριτική του καπιταλισμού από πλευράς της Γκουε. Καλά, το πούμε σε μια άλλη φορά. Τώρα, Όσον αφορά αυτή την έκθεση, συμβρούμε με τα περισσότερα που έγραψε η συγγήτρια και με τις περισσότερες τροπολογίες. Και για την 1 και για την 3 όμως να δούμε κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν με την αρχή της κοινή αγοράς. Γιατί υπάρχουν σε αντίκειτο σε διατάξεις για την δημοσίευση. Γιατί να μην ισχύουν αυτά και για τον ενιαίο μηχανισμό. Ναι, γιατί να μην αποκλείουμε από ό,τι είναι εφαρμοστεί ή τον υπόλοιπη γενιά Να το δούμε. Πέραν αυτού πάντως, κινούμαστε στο ίδιο μήκο σχήματος. Επίσης, προσέξαμε ότι συμφωνούμε πάνω κάτω με την τροπολογία μας 18 τρόσο να αφορά αυτού του είδους την ε, προθεσμία εκπνοής βέβαια θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία άσχετα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Άρα είναι θεμητό. Αυτές οι περίοδοι να επιδέχονται παράταση. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με την μέθοδο υπολογισμού όσον αφορά τα ημερήσια πρόστιμα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τα εφάπαξ και τόσο πολύπλοκα πρόστιμα. Όταν για θέματα υποπτικά έχουμε 730 730 ευρώ για την ε, ημερήσια, ενώ είναι 150 για τα υποπτικά. Ας βάλουμε απλώ τον υπολογισμό και το ίδιο ποσό. Τώρα όσον αφορά τις τροπολογίες συναδέλφων. Καταλαβαίνω τι προβληματίζει τον Μάρκο Φέρμπερ. Μα λέει βασικά θα πρέπει να υπάρχει δημοσίευση των ε, κυρώσεων πριν υπάρχει η, η ευκαιρία, η δυνατότητα τέλο πάντων κανεί να προσφύγει κατά τη επιβολή τη κύρωση. γιατί γιατί πώ να δημοσίευσει μια κύρωση αν κανεί δεν είναι βέβαιο. Μπορεί να γίνει ένα λάθο. Όλοι κάνουν λάθη, ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα. Άρα καταλαβαίνω πού το πάει στο 16 ο Μάρκος Φέρμπερ. Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσον υπάρχουν ε, κάποιου ε, όρια, προθεσμίες τέλο πάντων για την δημοσίευση. Ε, γιατί εδώ δεν, ε, δεν αποκλείεται να μην υπάρχει καθόλου δημοσίευση, γιατί έχουμε την κοινή αρχή του κοινωτικού δικαίου, ότι όλες οι κυρώσεις δημοσιεύονται. Άρα ίσως το πρέπει να βρούμε κάποια διατύπωση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε εδώ τη βασική αρχή. Αλλά να μην καταλήξουμε στο ότι ακριβώς λόγω της περίοδου ισχύω και εκνοής της διάρκειας, αν κανείς προσφύγει σε δικαστήριο, να αποφύγει την ε, δημοσίευση. Γιατί αν κατάλαβα καλά, δεν θέλει αυτό να προτείνει ο Μάρκος Φέρμπερ. Άλλωστε αυτό θα αντέβαινε με την αρχή του κοινωτικού ε, δικαίου για τη δημοσίευση. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε συμβασμό. Ε, δεν είναι εδώ πέρα, δεν πρόκειται για τη μεγάλη μας ε, διαφωνία όσον αφορά με την πάλη των τάξεων και τον καπιταλισμό. Μπάλτς, γιατί ζητείς το λόγο. Σύντομα. Θα ήθελα κι εγώ να πω από τη δική μου τη σκοπιά πως πράγματι είναι σημαντικό να πούμε πως θα γίνει η δημοσίευση μόνο όταν εξαλειφθούν όλα τα ε, ένδικα μέσα όσον αφορά τις ε, ποινές, αλλά κάτι άλλο είναι σημαντικό νομίζω δεδομένων και των ε, διεθνών εξελίξεων. Δεδομένων των όσων γίνονται και στις ΙΠΑ. Ε, Τους τελευταίους μήνες είχαμε κάποια παραδείγματα με αποτρεπτικό νομίζω χαρακτήρα θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για συνεργασία και συνεννόηση για μια πολιτική κυρώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρω πως δεν είναι απλό και ε, εντάξει, μπορεί να ακούγεται ως μια απλή έκκληση αλλά νομίζω πως θα πρέπει τελικά κάποιος ο οποίος ε, έχει κάνει κάτι, να, κάτι λάθος να πληρώσει κιόλας στο τέλος, έτσι. Είτε μιλάμε για θηγατρικές ε, ξένων εταιριών ή δικές μας ε, εκτός ε, Ευρώπης. Ε, πρέπει να δούμε όμως εδώ πέρα το να μην στερβλώνεται και ο ανταγωνισμός, γιατί πάρα πολλές ε, τέτοιες κυρώσεις νομίζω έφταναν στο σημείο να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε μια πολιτική κυρώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα και εγώ τέλος να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και βεβαίως ε, να στήριξω πλήρως τις προτάσεις και τις τροπολογίες του Μάρκους Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε αργήσει. Σύντομα κύριε γρήγορα πρόεδρε, ακούσαμε εδώ την πρόεδρο του Συμβουλίου Εποπτείας και είπε ότι θέλει εξευρωπαϊσμό της τραπεζικής αγοράς. Οπότε και έτσι να έχουμε καθαρά ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οργανισμούς. Όλοι συμφωνούμε γι' αυτό, αλλά βέβαια υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι ας πούμε το να μην υπάρχει αρκετά πρικοδοτημένο ταμείο πύλησης διαφόρων για όλη αυτή την περίοδο και επίσης να υπάρχει κάποιο είδου εξασφάλιση των καταθέσεων. Στην προηγούμενη θητεία η Οικονομική Επιτροπή έδωσε μάχες ούτως ώστε να πλησιωθεί σωστά οικονομικά το Ταμείο Πύλησης των Διαφορών. Ήρθε σε την παράθεση με το Συμβούλιο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ε, τραπεζικής αγοράς στη συνέχεια, συγγνώμη, τραπεζικής ένωσης συνέχεια και της αγοράς και να μπορέσει να επιβιώσει. Όποτε γι' αυτό φτάσαμε σε αυτές τις κυρώσεις αυτού του κανονισμού και του προηγούμενου, οπότε είπαμε ότι θα ισχύσουν όσο χρειάζεται για να έχει η Τραπεζική Ένωση την σκοπόμενη αξιοπιστία. Είπαμε επίσης ότι αυτά δεν είναι μόνο θέματα του, ε, του επίτροπου, αλλά όλα αυτά πάνε στον γενικό προπολογισμό. Θα πρέπει να έχει περιεχόμενη τραπεζική ένωση πάνω απ' όλα. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν αρκετοί πόροι για αυτό το Ταμείο Επίλυση Διαφόρων. Κέρι, έχεις το λόγο τώρα. Εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θα συζητήσω με όλους τους συζητητές τις επόμενες 24 ώρες να δούμε αν θα συμφωνήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Στα υπόλοιπα είναι σαφή, συμφωνούμε, λίγες οι διαφορές. Προτείνω λοιπόν να στείλω γραπτές συμβιβαστικές προτάσεις επόμενες 24 ώρες, να συνενεθώ και με τη γραμματεία, να δούμε εάν συμφωνούμε και αν βεβαίω είναι συμβατά με τα υπόλοιπα νομοθετήματα. Δεν είναι μόνο η οδηγία περί κεφαλιακής επάρκειας, αλλά και ο μηχανισμός σταθερότητας, ο ενιαίος οπτικός μηχανισμός και οι κανονισμοί κατάχρησης ε, δεσπόζουσας θέσης, ε, θα τα δούμε αυτά με την γραμματεία τις επόμενες 24 ώρες. Αυτά και ελπίζω και οι επόμενες εκθέσεις μου να είναι τόσο απλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο. Α, μου λένε εδώ πέρα πως η ψηφοφορία θα γίνει στις 11.11 του. Μαζί με την άλλη έκθεση για τα στατιστικά στοιχεία κανόνες για τη χρήση των στατιστικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, ε, το επόμενο θέμα είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013. Παμπλο Τζάλμπα Μπιντεγκάιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο θα πρέπει να σας πιω ποιο είναι το πλαίσιο του παιδιού μας αυτή την έκθεση. Πρόκειται για κάποια έκθεση του 2013 της Κεντρικής Τράπεζας αλλά είπαμε ότι όλα αυτά θα αρχής αρχής του 2014 που είχαμε κάποια σοβαρά γεγονότα στα πλαίσια της πορείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οπότε και είχαν ανακοινωθεί σημαντικά μέτρα όσον αφορά την συγκυρία του 2013. Είχαμε το ότι παρά το 0,4% την πτώση του ΕΛΚ και είχαμε 12% ανεργία. βλέπαμε επιτέλους φως στην άκρη του τούνελ οπότε και αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα δείγματα ανασυγκρότησης και αναθέρμανσης της οικονομίας κάτι το οποίο τελικά ε, ολοκληρώθηκε το 2014 οπότε και λένε διάφοροι ότι βρισκόμαστε πρώτων φυλών ε, άλλη, άλλη και ότι η οικονομία δεν προχωρεί όπως θα θέλαμε. Αλλά πάντως είναι θετικά τα δείγματα που σας είπα. Γι' αυτό και βλέπουμε 1,2 ως ε, ρυθμό ανάπτυξης για φέτος. Τώρα, όσον αφορά τον πληθυσμό του 2013, είχαμε πληθυσμό που έτρεχε στην Ευρωζώνη με 1,3% μακράν του στόχου που είχε τεθεί ε, από την Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή να είναι περίπου το 2% πληθωρισμός. Στο χαμηλότερο επίπεδο ήταν το 0,3% φέτος, πάλι πολύ μακριά από το στόχο που έθεσε η Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τις πιστώσεις, 2013, είχαμε αρνητικούς ρυθμούς πλην 2,4 της πιστώσης ιδιωτικού τομέα. Πλην 2,4. Και όπως είπαμε σήμερα και όσο μας παρουσίασε η, η πρόεδρος του Επιτικού Συμβουλίου είχαμε κατάτμιση των αγορών. Κάτι το οποίο ρίχνει τα, τις πιστώσεις. Συνεχή πτώση επομένω, αλλά επίσης έχουμε διαφορές μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου ή της ε, Βορείου Ευρώπης. Περισσότερο έχει πληγεί επομένω η περιφέρεια. Και άρα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την όθηση που προδοθεί στην ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόληση. Είναι αλήθεια ότι το 2013 θεωρήσαμε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να λάβει κάποια πιο αποτελεσματικά μέτρα. Για αυτή την κατάτμιση των χρηματαγόρων. Μας λείπουν επομένω τέτοια αποτελεσματικά μέτρα. Δεν έγινε το 2013. Οπότε θα πρέπει να πούμε μπράβο στην Κεντρική Τράπεζα γιατί αντέδρασε ακαριέα οπότε ανακούφισε τις χρηματαγορές και βοήθησε ούτως ώστε να ξαναγυρίσει η εμπιστοσύνη προς το ενιαίο νόμισμα. Γι' αυτό και είχαμε συρρήγνωση των επιτοκίων για χρηματοδότηση των κρατών μελών. Και επίση θα έπρεπε όσον αφορά τι πληρωμές για την ίδια τράπεζα να εισφέρουν λιγότερο τα κράτη-μέλη. Βέβαια πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι αυτή του είδου οικονομική ε, ανασυγκρότηση και η δημιουργία τη απασχόλησης απαιτεί κοινή δράση. Μόνο με νομισματική πολιτική δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Και μια τέτοια επικρατική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από μια καλύτερη εφαρμογή από τα απλώς των κρατών μελών της πολιτικής. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερη εφαρμογή από πλευράς των ε, Ευρωπαϊκών Δεσμικών Οργάνων. Να μην ξεγελιόμαστε, μην ξεγελούμε και τους πολίτες, ότι μόνο με νομισματική πολιτική θα δώσουμε όθηση σε ανάπτυξη και απασχόληση. Χρειάζεται κοινή δράση. Και έτσι να έχουμε εξελίξεις θετικές βιώσιμες. Τον Ιούνιο φέτο είχαμε κάποιες αποφάσεις και είπαμε πάμε σε επενδύσεις ενός δις και φτάνουμε έτσι σε επίπεδα αρχών 2012. Όλα αυτά τα μέτρα ήταν καλοδεχούμενα, αλλά έτσι απλώς κερδίσαμε χρόνο. Έτσι κερδίθηκε χρόνος για να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις τα κράτη-μέλη και να λάβουν και τα θεσμικά όργανα τις αναγκαίες αποφάσεις, ούτως ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε για την πολιτική ολοκλήρωση. Μόνο η Κεντρική Ένωση δεν μπορεί να λύσει τα διευθυντικά προβλήματα των κρατών μελών τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενεργήσουν. Και έτσι να υπάρξει μια στέρεη βάση, οπότε να πάμε για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωζώνη. Επεκτατική οικονομική πολιτική δεν μπορεί να τονώσει την ζήτηση. Τα μέτρα της και τράπεζας έχουν μεταβατικό χαρακτήρα. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δίνουν χρόνο στα κράτη-μέλη και στα θεσμικά όργανα. Τόσο ώστε να μπορέσουν να εξηγιάνουν τα δημοσιονομικά του και να κάνουν τι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Να υπάρχουν οι κατάλληλε συνθήκε για να δημιουργηθεί ανάπτυξη και απασχόληση. Επίση πρέπει να πούμε ότι η Ευρική Κέντρια Τράπεζα τελείωσε ανεξάρτητα χαρές νομισματική πολιτική. Ακριβώ, όπω τάσουν οι συνθήκε επίση θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε τον ε, πρώτο πυλώνα της ε, Νομισματικής Ένωσης, έχουμε τον μηχανισμό της ε, το που θα αρχίσει να τρέχει από αύριο, 4 Νοεμβρίου. Και να έχουμε ένα ενιαίο εργοτικό σύνδεμα στην Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλο βήμα. Οπότε τώρα θα έχουμε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και σταθερότητα. Εν κατακλείδη σας υπενθυμίζω ότι η εποπτεία και του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο ώστε να έχει αξιοπιστία ο μηχανισμός της εποπτείας. Αυτά για την εκθεσή μου και βεβαίως είμαι τώρα στη διάθεσή σας εάν κάτι θέλουν οι συνάδελφοι ή κυρίως βέβαια οι σκιώδεις συνεισηγητές. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Λόγω τώρα στους κοιόδης εισηγητές. Θα ζητήσω τους, από τους συναδελφούς να μιλήσουν για ένα τρίλεπτο. Διότι δεν έχουμε πλέον πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ο κ. Σόλου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. δεν έχουμε συναντηθεί ακόμη. Ήδη θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο αυτή την εβδομάδα, οπότε στην επόμενη και μόνο συνεδρία θα μπορέσω να τοποθετηθώ το σχετικά. Ευχαριστώ για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, να πούμε ότι Πρόκειται ουσιαστικά για μια τοποθέτηση επί μιας εκθέσεως 300 σελίδων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και νομίζω ότι τα θέματα που έχει θίξει, ότι υπάρχει υποτονική ανάπτυξη, ε, ότι είχαμε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και για το 2013, πράγματι ισχύουν. Απλά πρέπει να μιλήσουμε για μια ανάπτυξη η οποία όμως να δημιουργεί θέσεις εργασίας και όχι γενικώ να υπάρχει μια ανάπτυξη στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για το χτύπημα της ανεργίας η οποία πραγματικά έχει φτάσει σε εφιαλτικά σημεία ιδίω για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου γιατί υπάρχει μια απόκληση στα ποσοστά ανεργίας από 5 έως 26%. Και αν πάμε στην ανεργία των νέων, στην Ισπανία είναι 53,7%, στην Ελλάδα 50,7%, στη Γερμανία όμως 7,6%, 9% στην Αυστρία. Τα θέματα λοιπόν είναι σοβαρά, όπως επίσης και το ζήτημα του αποπληθωρισμού, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως επίσης και το ζήτημα της ρευστότητα, διότι είναι δεδομένο ότι παρότι οι τράπεζες χρηματοδοτήθηκαν με ε, πάνω από 1,6-3 εκατομμύρια ευρώ, ε, τελικά ε, δεν έριξαν αυτά τα ποσά στην ίδια την αγορά. Θέλω όμως να θίξω ένα θέμα για τον εισηγητή για να το έχει υπόψη για την, ε, όταν συναντηθούμε. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που σωστά έχει τεθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και το άρθρο 123 δεν μπορεί να χρηματοδοτεί κυβερνήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει στο άλλο άκρο. Διότι αν δείτε τα ποσοστά και τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το 2013 είχε κέρδη 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 961 εκατομμύρια ευρώ τα έχει από τα ομόλογα, τα οποία έχει αγοράσει των κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου κυρίως από τη δευτερογενή αγορά. Και αυτά τα ομόλογα τα έχει αγοράσει με έκπτωση τουλάχιστον 40%. Έβγαλε λοιπόν κέρδος 961 εκατομμύρια ευρώ για το 2013, εκ των οποίων 437 εκατομμύρια ευρώ κέρδος μόνο από τα ελληνικά ομόλογα. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι αδύνατον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει ομόλογα με έκπτωση τουλάχιστον 40% και να ζητά να τα πληρώνεται στην ονομαστική τους αξία. Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα ότι φέτος θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πληρώσει μόνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το ποσό, την υπερβάλλουσα διαφορά, για μένα είναι ξεκάθαρη κερδοσκοπία. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίζει αυτή τη δουλειά να την κάνει η Κεντρική Τράπεζα. Αν δείτε τα ποσά μάλιστα που έχει η Κεντρική Τράπεζα, ο κέρδη είναι στη σελίδα 225 της έκθεσής της, και στη σελίδα 100 της έκθεσής της μπορείτε να δείτε ότι αυτή τη στιγμή έχει ομόλογα αξίας 180 δισεκατομμυρίων ευρώ που τα αγόρασε στη δευτερογενή αγορά. Η πρότασή μας λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πληρωθεί το ποσό το οποίο έδωσε για να αγοράσει αυτά τα ομόλογα, υποτίθεται για να βοηθήσει τα κράτη και για να στηρίξει το ευρώ και να πάρει ένα επιτόκιο το οποίο σήμερα είναι 0,15% δεν μπορεί να βγάζει αυτά τα υπερβάλλοντα κέρδη. Επομένω και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε γιατί θα δώσω στοιχεία στον εισηγητή στο θέμα αυτό γιατί για μα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε η αντίληψη που λέει η Κεντρική Τράπεζα θα σα δώσω την επόμενη χρονιά τα κέρδη ισχύει. Πρώτον, διότι για να πληρώσει σήμερα η Ελλάδα ένα ομόλογο τη Κεντρική Τράπεζα 10 δισεκατομμύρια ευρώ αναγκάζεται να δανειστεί από τον ESM, αναγκάζεται να δανειστεί από το ΔΝΤ για να πληρώσει φέτος στην ονομαστική του αξία αυτό το ομόλογο και να πάρει, αν θα πάρει του χρόνου, πίσω ορισμένα κέρδη, τα οποία μέχρι στιγμής δεν τις δίδονται. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κράτη. Επομένως αυτό το σημείο πρέπει να το συζητήσουμε αναλυτικά, να έχουμε την ευκαιρία σε μια άλλη συνεδρίαση να θέσουμε όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσει ανάσα στα κράτη-μέλη, διότι τα ομόλογα Τις τράπεζες πρέπει να πληρωθούν στην αξία που τα αγόρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι στην ονομαστική τους αξία, κερδοσκοπώντας έτσι εις βάρος των κρατών, εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους φιλελεύθερους, ο κ. Ε, Ραμόν Τρεμόζα Μπάλτσεφ που δεν είναι εδώ ε, για τους φιλελεύθερους. Περνάμε στην ΚΟΕ. Ναι. Αλλά θα είμαι πολύ πιο σύντομη γιατί τα είχα πει αυτά που ήθελα να πω. Να ζητήσω συγγνώμη από τη γραμματεία. Διότι δεν πληροφόρησα ότι δεν θα μπορούσα να συμμετέχω στην ε, ε συζήτηση για τις κυρώσεις. Και είχα άλλη συζήτηση σε άλλη επιτροπή, γι' αυτό έγινε αυτό το μπέρδεμα. Τέλος πάντων συμμετείχα χωρίς να το γνωρίσω. Πολύ γενικό σχόλιο, ήδη τα είπα προλίγου. Νομίζω ότι ο Πάμπλο ήταν εδώ, τα άκουσε. Είμαι, δεν είμαι σκιώδης συγκεντρία της ΓΚΟΕ, αλλά Κάποια από τα εισαγωγικά σχόλια του Πάμπλο έχουν θεμελιώδη σημασία και για μα. Καταλαβαίνω ότι για την ανάλυση των δραστηριοτήτων του ε, τη ΕΚΤ δεν θα έχουμε και απόλυτη σύγκληση απόψεων μεταξύ μα. Όμω, όπω υπόσχε και προ θα πρέπει να δούμε την νομισματική πολιτική και τι επιπτώσει του, να δούμε τι αποτυχίε τη. Απλώ να μην περιοριζόμαστε στο να θριαμβολογούμε για τα θετικά αποτελέσματα και προ το ρόλο του Κοινοβουλίου πρέπει να κάνουμε κάποιες συστάσεις. Όπως το λέμε συχνά, ε, πρέπει να υπάρξει ένα πώληση μίξ, τα είπα και πριν. Ιδάλω δεν μπορεί η νομισματική πολιτική να είναι αποτελεσματική και να μας βγάλει από την κρίση. Γιατί οι πολιτικές λιτότητας σκοτώνουν κάθε πρόθεση ε, μια σωστή νομισματικής πολιτικής. Οπότε οι επενδύσεις εδώ έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο. Και το δεύτερο στοιχείο, κάτι που το ε, στη σχολίασε και ο Πάμπλο, ότι δηλαδή η ιδιαίτερα επεκτατική νομισματική πολιτική δεν επιλύει τίποτα χωρίς χρήμα που να φτάνει στην πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα, δεν μπορεί το χρήμα να μην φτάνει στην πραγματική οικονομία εάν δεν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες για να διευκολυνθούν. Θα πρέπει λοιπόν, ε, εάν δεν τροφοδοτήσουμε τις τράπεζες με χρήμα, που να πηγαίνει στην πραγματική οικονομία, να περιμένουμε την κερδοσκοπία τους. Δεν φτάνει η λογιστική λογιστικίστικη αντιμετώπιση των ισοζυγίων των τραπεζών για να φανεί ότι υπάρχουν τα απαραίτητα ποσά. Πρέπει να φτάσουν και στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους, ο κ. Ουρτασούν. Τρεις βασικές ιδέες και κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα, πρέπει να τονίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ενεργήσαμε με βραδίδιτα πολύ πιο ταχύως θα έπρεπε να αναλάβουμε δράση. Επίσης, δεν λέει το κείμενο ότι από πλευράς τιμολογιακή πολιτικής δεν κάνει τη δουλειά της η κεντρική τράπεζα. Ενώ έχει εντολή προς τούτο. Άλλο. Τρίτο. Η έκθεση θέλει να καλύψει. Αυτό που είπε ο Τζάξον Χόλο πρόεδρος, δηλαδή πώς θα συνδυάσουμε την πολιτική της ε, Κεντρικής Τράπεζας από πλευράς αύξησης της ζήτησης. Έχει δίκιο η Μαλίσσα Ματίας. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση γιατί ε, η παίκτης 2013 δεν, ε, δεν, δεν καλύπτει τι έκανε, τι δεν έκανε γιατί τόσο αργά ενήργησε η Κεντρική Τράπεζα και το 2012 με την, ε, ε, την ε, Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία τέλο πάντων. Και οπότε και τώρα θα πρέπει να δούμε εκτός του τι έγινε, τι δεν έγινε. Είχαμε αυτή την επεκτατική πολιτική και το κάναν και άλλες τράπεζες. Τι έγινε όσον αφορά το κρατικό χρέος. Πόσο κόστησε αυτή η πολιτική στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω του ότι δεν έκανε αυτό που έπρεπε η Κεντρική Τράπεζα στον αφορά τον πιστωτή τελευταίας καταφυγής όπως λέγεται. Και εμάς μας κατέθεσε ο εθνικό προπολογισμό σαν Ισπανία. Τι έγινε με τον ε, προϋπολογισμό τι έγινε με αυτήν την ε, επικρατική νομισματική πολιτική. Δεν είχαμε τα κίνητρα από πλευρά Κεντρικής Τράπεζα. Άρα θα πρέπει τώρα να αποσύρει αυτά τα οποία έχει κάνει και ακόμα μερικά πράγματα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους νομικούς περιορισμούς. Φυσικά και φταίει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Πάντως, πάρα πολλά από τα έκτακτα μέτρα που πήρε η Τράπεζα μέχρι και αντιβαίνουν το κοινοτικού δικαίου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατισμός και έλεγχος επί της τράπεζας. Δεν υπάρχει τώρα, είναι ανεπαρκή ο έλεγχο. Σωστό είναι να δημοσιεύονται τα πρακτικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Όπω εδώ να δημοσιεύουν τις εκθέσεις. Ανεξαρτησία, τι θα πει. Πάει και από τη μία μεριά και από την άλλη. Όλα αυτά έχουν ε, μείνει στα λόγια, η ανεξαρτησία δηλαδή. Πού είναι εξαρτησία στις πράξεις και συγκεκριμένα στι διαρθωτικέ μεταρρυθμίσει ούτε στην αγορά εργασία έχουν ε, Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο έγινε. Τι έγινε με αυτή την περίφημη επιστολή Τρισέ προς τον Θαπατέρ. Όλοι ξέρουν. Αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν με την ε, κοινωνική τραπεζά. Δεν είναι δουλειά της. Τελευταίο τώρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι το έλασον κακόν τα, σχετικά με την εποπτεία. Έχουμε το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Θα πρέπει η, εποπτική αρχή να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Το λένε οι συνθήκες, αλλά εμείς θα το ζητάμε να ισχύσει στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριο Σόρο, θέλει λίγο το λόγο. Ναι, ε, Πρόεδρε, μετά το Στρασβούργο και τη Σύνοδο δεν τα συζητήσαμε με τους συναδέλφους και ήθελα απλώς να έχω τη δυνατότητα να τα πληροφορηθώ καλύτερα. Αλλά Και σε σχέση με την όλη συζήτηση που μόλις έγινε και όσα θα είχα εγώ να πω προκαταρκτικά, θα ήθελα να τοποθετηθώ τελικά. Λοιπόν, για τον εισηγητή χαίρομαι από το σημείο, για το σημείο αφετηρίας του, ε, πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση και τις κοινωνικές παραμέτρους, την, ε, τα φοβερά επίπεδα ανεργία σε ορισμένες χώρες, που είναι ένα σημείο κλειδί, και το ότι όλοι πρέπει ε, από κοινού να ενεργοποιηθούμε. Κοινωνικοί παράγοντες λοιπόν, ενεργεία ενεργεια των νέων, ανάπτυξη, εξή σε ορισμένες χώρες με αύξηση του επίπεδου φτώχειας, χώρας ε, που ξεπερνά το 25% ε, των οικογενειών που βρίσκονται σε συνθήκες σχετικής ένδυας. Συμφωνώ ότι η νομισματική πολιτική απομονή δεν μπορεί να εξισορροπήσει την κατάσταση. θα πρέπει κάπως να ξαναπάρει μπρο αυτή η Ευρώπη μας, ιδίως σε κάποιες χώρες. Ωστόσο, Εφόσον δεν φτάνουν νομισματικές πολιτικές, πρέπει να αναζητήσουμε συμπληρωματικές πολιτικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις μόνον στις επιμέρους χώρες είναι οι πολιτικές που μας λείπουν, ούτε οι δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά και οι δημοσιονομικές πολιτικές, εφόσον αποδυναμώνονται ε, μαζί με την κυριαρχία των επιμέρους χωρών, που καλούνται να συμμορφωθούν με το σύμφωνο σταθερότητας, με το δημοσιονομικό όπως ονομάστηκε σύμφωνο. Και δεν μπορούν με το έλλειμμα τους να χρηματοδοτήσουν πλέον μεγάλες πολιτικές ε, επενδύσεων, για να ξαναρχίσει η ζήτηση, για να υπάρξει περισσότερη απασχόληση. Κάποιο πρέπει επιτέλου να ξαναπυροδοτήσει αυτέ τι επενδύσει. Ένα σημαντικό στοιχείο που επανέρχεται στι συζητήσει μα, ιδίω με τον κύριο Γιουνκέρ, είναι ότι ζητούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων, μεγάλων ευρωπαϊκών επενδύσεων, 35 δι ευρώ για τα ερχόμενα 5 χρόνια. Ακόμη και αν ε, προ μεγάλη μα έκπληξη είπε πρόσφατα ο κύριο Γιουνκέρ στο Στρασβούργο ότι αυτέ οι νέε μεγάλε επενδύσει θα πρέπει να έρθουν χωρίς χρέος και διερωτώ πώς, πώς, λες και θα κληθούν οι ιδιώτες να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, τέλος πάντων, έτσι δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωρήσουμε. Υπάρχει ανάγκη να προωθήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων για να υπάρξει ανατέρμανση τη ζήτηση και δημιουργία αναθέσεων εργασία. Μάλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που προσφάτω ανέλαβε τη δέσμευση σε μεγάλο βαθμό να αλλάξει τα μεταβλητά ομόλογα ε, θα μπορούσε ενδεχομένως να αγοράσει τίτλους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έτσι να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ευρωπαϊκών, ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κληθεί να χαράξει καινοτόμε πολιτικέ για να υπάρξει ένα θέρμανση τη ζήτηση. Αλλά η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει μόνο με τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει τη επιμέρου χώρε. Και συμφωνώ και εγώ με τον συνάδελφό μου, με τον προηγούμενο συνάδελφο, ότι στο σημείο 16 στο σημείο 16 του ε, σχεδίου έκθεσης δεν πείθομαι, δεν πείθομαι ούτε εγώ ότι η νομοσματική πολιτική φτάνει και ότι φτάνει μόνο η... Η νομισματική πολιτική που διευκολύνει θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με... και ότι φτάνει η ποσοτική χαλάρωση. Το ίδιο που γίνεται στις ΗΠΑ θα πρέπει να το δούμε και εμείς. Ε, και το συζήτησα πρόσφατα για με κάποιο συνάδελφο. Η Bundesbank εξέδωσε κρατικά ομόλογα 39 ε, χρόνων με 2% Τόκιο, Άρα τα ερχόμενα χρόνια θα δούμε επίπεδα ε, ε, αύξηση των δανείων πολύ χαμηλά και πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης γενικότερα αλλά και τέτοιε διάρκειες τα ομόλογα, 31-32 χρόνια. Σε τέτοιου είδου συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να ανησυχήσουμε πολύ περισσότερο και να σκεφτούμε πώς θα ενεργοποιήσουμε μηχανισμούς ανάπτυξης, ακόμα και με μη συμβατικά συστήματα που ξεφεύγουν από την κλασική σύνεση με την οποία άκουσα να τοποθετούνται κάποιοι ε, αυτούς τους πρώτους μήνες τη Βρυξέλλες. Ε, τέλος, Πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε και άλλο ένα θέμα που το συζητούν πολλοί οικονομολόγοι στην Ευρώπη, ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει ως αρμοδιότητα την νομισματική πολιτική και τη σταθεροποίηση του επίπεδου των τιμών, αλλά και των ε, ε, επιτοκίων, Α δούμε σε σύγκριση με αυτό τι γίνεται στι ΗΠΑ, μια άλλη χώρα με τι οποίε έχουμε πολλέ ε, οικονομικέ συναλλαγέ έχουμε ε, μειωμένη δυνατότητα ανταγωνισμού ε, λόγω αυτών των ε, χαμηλών επιπέδων. Και τέλος, μιλάμε για 18 χώρες. Έχουμε στην Ευρωζώνη ένα κοινό συντελεστή. Όμως, με αυτό το συντελεστή με την κοινή αυτή ε, ε τιμή του ευρώ 1,21 πόσο είναι ακριβώς σήμερα αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες χώρες που είναι πολύ ανταγωνιστικές είναι πολύ μικρή τιμή ενώ για κάποιους άλλους είναι πολύ υψηλή χώρες που είναι λιγότερα ανταγωνιστικές Πώς λοιπόν θα συγκλίνουμε εφόσον δεν έχουμε κανόνες σύγκλησης ε, με το ενιαίο νομισματικό σύστημα που ε, κατέρευσε το 1992. Εκεί υπήρχαν κάποιες λύσεις. Αλλιώς ο μόνος μηχανισμός σύγκλησης που έχουμε είναι η εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή αύξηση της φτώχειας σε ορισμένες χώρες εις βάρος κάποιων άλλων χωρών που γίνονται πλουσιότερες. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Εκεί πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε στη συνέχεια τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πώς θα συνδυάσουμε τόσε οικονομίε, 18 οικονομίε που μαζί φαίνεται ότι τελικά δεν συμβαδίζουν. Υπάρχει ανάγκη σύγκληση. Διότι η ένδυα και η οδήγηση στη φτώχεια ολόκληρων χωρών και περιοχών της Ευρώπης, ολόκληρων ομάδων πληθυσμού, δεν είναι ε, λύση αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ως προβληματισμό στα θεμέλια της σύνταξη της έκθεσής μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόρου και τώρα ο εισηγητής. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς κύριε Πρόεδρε για τα όσα ε, πρότειναν. Και τώρα επιτρέψτε μου να πω κάτι πρώτα για τον κύριο Σόρου, τον σοσιαλιστή συνάδελφο. Πρώτα πρώτα δεν είπε κανείς ότι το μόνο το πρέπει να γίνει είναι νομισματικές πολιτικές για να έχουμε απασχόληση για να δεις ναι, ναι, ναι, όπως το είπατε, χρειάζεται πρόγραμμα επενδύσεων, ισχύει. Και όπως επίσης και κάποιες χώρες οι οποίες είναι σε θέση να μπορέσουν να κάνουν ε, πιο επεκτατική δημιουργική πολιτική, μπορούν να το κάνουν αυτά, αλλά επίσης τα είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανειλημμένα εδώ, είστε κατά, αλλά όπως είπε και η Μαρίσα Ματίας, είναι σημαντικό το policy mix. Και φυσικά policy mix δεν μπορεί να πει μόνο νομισματικές, ε, μόνο νομισματική πολιτική, μόνο τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Το, το είπαν και άλλοι, δώσα από τον υπόλοιπο. τώρα, για το σημείο 16, κοιτάξτε τι λέει, για τα κίνητρα. Δεν πρέπει να παρεμεθεί αυτό. Αλλά επίσης δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον θεωρώντας ότι τα μέτρα, τα μη συμβατικά, τα κινήτρα, όλα αυτά ότι, ότι, ότι είναι ανεξάντλητα. Χρειάζονται μέτρα έχοντας υπόψη ότι όλα έχουν κάποιο όριο. Προσοχή να μην φτάσουμε και να γίνει μπούμεραγκ αυτό. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι να βρει τη σωστή ισορροπία κινητική Κεντρική Τράπεζα μεταξύ του κινδύνου της πρόορης εγκατάλειψης της νομισματικής πολιτικής και από την άλλη μεριά των κινδύνων που έχουν ε, ε, σχέση με αυτήν την εγκατάλειψη, με αυτή την στροφή. Πρόορη αλλαγή. με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και έχοντας υπόψη κάποια τυχόν δυσμενή αποτελέσματα. Ο κύριος Μαριάς τώρα. Συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο με τέτοιου ε, ε, στοιχεία θετικά ε, δεν, δεν, αρκεί ε, για να κατέβουμε συμπεράσματα χρειάζεται να δούμε και στοιχεία από την απασχόληση. Το έχουμε πει αυτό επανειλημμένα και ακριβώ δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ακριβώ η δημιουργία τη απασχόληση μπορεί να προέλθει μόνο και αποκλειστικά από μια νομισματική πολιτική. Όμω αυτό ε, θεωρώ ότι δεν είναι από μόνο το αρκετό. Δεν θα πρέπει να το βλέπουμε απομονωμένα το θέμα. Κυρία Μαρία, επίση συμφωνώ μαζί σα και όπω προείπα είναι σημαντικό το τι πόληση μίξ έχουμε και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να φτάσουμε σε μια ανάπτυξη όχι μόνο νομισματικά. Και γι' αυτό στην έκθεση αναδεικνύουμε το πόσο σημαντικό είναι τούτο. Τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος από τους πράσινους ε, ότι έκανε λάθη και αντέδρασε αργά και η τράπεζα. Όμως αυτό γιατί έγινε. Γιατί όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι και εκείνοι δεν έκαναν ό,τι έπρεπε και όταν έπρεπε έκαναν τα λάθος πράγματα και τα κάνανε και αργά. Κάνει ό,τι μπορεί στα πλαίσια εντολής τη η Κεντρική Τράπεζα που κινείται στα πλαίσια των συνθήκων. Ε, Επίση, είπαμε και για τον πληθωρισμό και γι' αυτό ισχύει το ίδιο, αυτό που σας είπα, κύριο Τασούν, Τώρα έχουμε για τα σημεία 15 και 16. Τα ξεκαθαρίσαμε, αν θέλετε. Νομίζω πίσω ότι σας κάλυψα και για τα περισσότερα βασικά. Ευχαρίστως και σε συνεδρίαση και εκτός συνεδρίασης να ακούσω τη γνώμη σας για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να διαμορφώσουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση για τους στόχους που έχουμε τάξει να πετύχουμε. Ευχαριστούμε. Οπότε νομίζω μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη αυτής της συνεδρίασης. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή των απολογιών είναι 11 Νοεμβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου και την ίδια ημέρα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση και θα συναντηθούμε αύριο το πρωί. Με ψηφοφορία θα ξεκινήσουμε. Ψηφοφορία παρακαλώ να είστε όλοι εδώ στην ώρα σας.